Λοιπόν, παρακαλώ καθίστε. We continue with the meeting. Συνεχίζει η συνεδρίασή μας. Καθίστε παρακαλώ. Καλημέρα σε όσους ήρθανε, τους βουλευτές. Α, ο κύριος Ρωμέβα είναι ο μόνος βουλευτής ο οποίος ήρθε. Συνεχίζουμε με την ημερησία διάταξη που προβλέπει το σεμινάριο για τη μεταρρύθμιση της αλληλευτικής πολιτικής για τη Μεσόγειο και τον εύξηνο πόντο. Ε, καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ και να χαιρετήσω όλους αυτούς που είναι παρόντες να συγχαρώ τους εισηγητές οι οποίοι έχουν επιληφθεί αυτού του θέματος που είναι μεγάλη σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας παρουσιάζω τώρα τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα λάβουν το λόγο. Ο καθηγητής Μάσιμο Σπανιόλο, ο οποίος είναι επικεφαλής του Ιδρύματος για την έρευνα στην Αλία και την Ικτιοκαλλιέργεια στο Σαλέρνο της Ιταλίας. Μετά ο καθηγητής ε, Χουάν Λουίς Σουάρες Τεβιβέρο, από το Πανεπιστήμιο της Σεβίλης για τη συνεργασία στα θέματα αλίας στη Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα και τέλος ο Δόκτωρ Κάντι, ο οποίος είναι ιδιωτικός σύμβουλος και ήταν πρώην τεχνικός γραμματέας στο ΦΑΟ για τα θέματα αλίας. Ξέρετε πάνω κάτω ποια είναι η διαδικασία για την ακρόαση, όπως ήθιστε. Θα δώσουμε το λόγο στους ε, ομιλητές για 15-20 λεπτά για να παρουσιάσουν το θέμα τους και στη συνέχεια οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα σε ένα διάστημα περίπου μιας ώρας. Έχουμε καθυστερήσει λιγάκι, γι' αυτό σας παρακαλώ να προσαρμοστούμε στο χρονικό περιθώριο για να μπορέσουμε να κλείσουμε εγκαίρως στις 12.30. Και δίνω τώρα το λόγο στον καθηγητή Σπανιόλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να συνοψίσω αυτή την αλληλευτική πολιτική στη Μεσόγειο στα λίγα λεφτά που έχω στη διάθεσή μου. Πιστεύω θα συμφωνείτε ότι δεν είναι εύκολο έργο αυτό και γι' αυτό προτιμώ να μιλήσω στα Ιταλικά. Η παρέμβασή μου θα προσπαθήσει να εξετάσει και να αναλύσει πιο συγκεκριμένα τις πτυχές της αλληλευτικής πολιτικής σε συνάρτηση με την ε, τροποποίηση που προτείνεται να εισαχθούν ε, εδαφικές, εδαφικά δικαιώματα χρήση στη Μεσόγειο μέσω μιας κατανομής ποσοστώσεων προσπαθίας και αλίες και αλλιεύματος. Ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καθορισμό ορίων ε, δαφικών με μια κατανομή ποσοστώσεων αλλιευμάτων, αλλιευμάτων και προσπαθίες αλλιευτικής. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι αφορά τον ορισμό των μέσων που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από την έποψη την επιχειρησιακή. Αυτή η τροποποίηση αφορά, δημιουργεί και διάφορα ερωτήματα για τους λόγους που προανέφερα. Πάνω απ' όλα ε, αυτό το σύστημα δικαιωμάτων ε, χρήσεως περιοχών μπορεί να ταιριάξει με την κατανομή των δικαιωμάτων μέσω της αγωγής κανόνων που αποφασίζονται από κεντρική αρχή διαχείρισης ή ένα δικαίωμα τέτοιο εδαφικό περιοχής μπορεί να χαρακτηριστεί περισσότερο από κανόνες που αποφασίζονται από τους ίδιους τους ε, εμπορευομένους. Αν λοιπόν θα έπρεπε να προβλέψουμε ότι η ζώνη είναι αντικείμενο κάποιας τέτοιας ποσόστοσης, το TERF δηλαδή αυτή η περιοχή, προέρχεται από κεντρικές αποφάσεις, διερωτώμεθα κατά πόσο πρόκειται περί TERF ή περί αδείας αλλιευτικής ειδικής που ήδη έχουμε στους κανονισμούς και στις υφιστάμενες διατάξεις. Τρίτο σημείο, τρίτο ερώτημα αφορά τα εδαφικά όρια και οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνουν ένα περιορισμό των δραστηριοτήτων στα ε, χωρικά ύδατα. Ε, δεν είναι πάντα αυτό ε, απαραίτητο. Απ' την άλλη πλευρά αυτό το σύστημα που προτείνεται είναι δυνατόν να μειώσει την υπεραλίευση και να συμβάλλει συνεπώς σε μια βιώσιμη σχέση μεταξύ πόρων ε, και αλληλευτικής προσπαθίας. Ή είναι δύσκολο να επιτευχθεί ο λόγω στόχος. Επιτρέψτε μου μια τάχιστη εισαγωγή όσον αφορά τα δικαιώματα χρήση. Τα δικαιώματα χρήση είναι σε δύο κατηγορίε. Δικαιώματα χρήση όσον αφορά του πόρου και όσον αφορά ε, τα χωρικά έδατα. Τα δικαιώματα χρήσεω των πόρων αφορούν ε, ποσοστώσει αλλιευμάτων, ε, δικαιώματα, ε, ποσοστώσει αλλιευτική προσπάθεια και μπορούμε να έχουμε δικαιώματα χρήσεως των πόρων που να είναι μεταφερόμενα. Αυτή η δυνατότητα μεταφοράς ε, δημιουργεί διάφορα προβλήματα τα οποία δεν θα εξεταστούν σε αυτό το πλαίσιο προφανώς αλλά όμως αντιπροσωπεύουν ε, μία πτυχή τεράστιας εμβελίας και σημασίας διότι με τη δυνατότητα μεταφοράς ε, οδηγούμεθα σε ένα σύστημα που ελέγχεται από κανόνες της αγοράς χωρίς τη δυνατότητα μεταφοράς. Η δημόσια, ο δημόσιος φορέας διαχείρισης έχει την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση. Σε περίπτωση όμως δικαιωμάτων, ε, εδαφικών δικαιωμάτων, ε, έχουμε υψηλό επίπεδο διαχείρισης ή συνδιαχείρισης, όπου η διαφορά εξαρτάται από το επίπεδο ε, εξουσίας που έχουν οι διάφορες οργανώσεις των αλλίων. Στον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, θα προσπαθήσω να δώσω κάποια παραδείγματα όσον αφορά τα δικαιώματα εδαφικά που υπάρχουν στη Μεσόγειο. Δεν υπάρχει ένα σχήμα που να ισχύει, ένα σχέδιο που να ισχύει για όλες τις καταστάσεις. Σήμερα έχουμε τέσσερα υποδείγματα που είναι το Κοφραντία στην Ισπανία, Προνταμή στην Γαλλία, ε, στα Στρακοειδή στην Αδριατική και τα διάφορα κονσόρτσια ε, βιοτεχνικής αλίας ε, που, που υπάρχουν στην Ιταλία. Ε, αυτά είναι τα μεγαλύτερα παραδείγματα που υπάρχουν. Θα δείτε όσο προχωρούμε με την όλη παρουσίαση ότι υπάρχουν και μεγάλες διαφορές μεταξύ των διαφόρων αυτών φορέων, των TERF όπως αποκαλούνται των ιστορικών, όπως της Κοφραντίας και την Πλυντομή, ε, και υπάρχουν και άλλα που βασίζονται σχέδιο διαχείρισης όπως είναι η Κοτζέμα και η Κοτζέμπα ένα χαρακτηριστικό κοινό όλων αυτών των παραδειγμάτων είναι ότι τα δικαιώματα αδερφής χρήσεως χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση εραστεχνικής παράκτειας ε, αλίας, κοντά στις ακτές δηλαδή. Άλλο χαρακτηριστικό που έχουν όλα αυτά που σας παρουσιάζω τα παραδείγματα είναι περιπτώσεις όπου οι κατηγορίες των αλλιέων ή των ενώσεων των αλλιέων των συνεταιρισμών αλλιέων μπορούν να καθορίσουν τους κανόνες της διαχείρισής τους. Αυτό ε, αληθεύει περισσότερο στην Κοτζέμο και στην Κοτζέμπα και δεν ισχύει τόσο στην Κοφραντίας και στην Πριντομή. Κάποτε ήταν έτσι τα πράγματα, τώρα έχει αλλάξει όμως η κατάσταση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, τα βασικά ενός τέρφ. Πρώτα απ' όλα το δικαίωμα καθορισμού της ε, περιοχής, του, της έκτασης. Οι ίδιοι οι εμπορευόμενοι το καθορίζουν. Δεν είναι κάποιος που το εξωτερικό ε, καθορίζει την περιοχή αλίας. Ε, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή, αυτός ο συνεταιρισμός ε, των αλλιών που θα καθορίσει ένα τόρφ έχει την εξουσία να καθορίσει και να εφαρμόσει τους κανόνες και αυτό είναι το χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί ένα τερφ από άλλα συστήματα διαχείρισης. Άλλο σημείο σημαντικό αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι εξωτερικοί φορείς μπορούν να συμμετάσχουν στην δράση που υλοποιείται από ένα TARF, δηλαδή να συμμετάσχουν σε ένα TARF, πώς μπορεί να καθοριστεί αυτός ο τρόπο συμμετοχή, με ποιο τρόπο μπορούν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους οι συνεταιρισμοί και ποιο είναι το επίπεδο των κινήτρων που απαιτούνται εντός ενός TARF. Αυτά εντάχει θα προσπαθήσω να σας τα περιγράψω. Ε, διότι όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Είναι σαφές ότι στην περίπτωση του καθορισμού της περιοχής Αλίας, τα δύο παραδείγματα ιστορικά, η Κοφραντίας και η Προυντομή, ε, δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης ε, μεγάλης, αλλά πρέπει να καταλάβουμε τις ρίζες της προσέγγισης που ακολουθούν. Έχουν διοικητικά όρια Δηλαδή, στην Κοφραντίας έχουν διοικητικά όρια που προέρχονται από το 12ο αιώνα όταν υπήρχε διαπραγμάτευση μεταξύ του, της Βασιλείας και των εκπροσώπων των Αλίων και καθόρισαν τα όρια. Οπότε είναι διοικητική φύσεω τα όρια. Δεν είναι τυχαίο και είναι πολύ ενδιαφέρον να καταλάβουμε το λόγο αυτόν, διότι μόλι ε, πρόσφατα αυτά τα διοικητικά όρια, αυτά τα χωρικά όρια ε, μεταφέρθηκαν σε μια διάταξη. Διότι μέχρι, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, εκ των πραγμάτων, το όριο ήταν de facto, αλλά δεν ήταν όριο νομικά κατοχυρωμένο. Τώρα όσον αφορά τους συνεταιρισμού για τη διαχείριση των ε, οστράκων, έχουμε ε, το top-down, ο περιορισμό top-down εκ των άνω προς τα κάτω όσον αφορά ε, τα μύδια. Τα όρια ακολουθούν προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή το κράτος καθορίζει τα όρια, οπότε υπάρχουν ευθύνε ακριβείς που καθορίζονται. Όσον αφορά την κοτσέπα, και την ε, ερασιτεχνική αλληλεία ε, υπάρχει αντίθετα. τη βιοτεχνική αλληλεία. Ακολουθούμε από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση. Οι ίδιες οι κοινότητες των αλληλείων καθορίζουν τα όρια ε, του χώρου αλληλείας των συμφερόντων τους. Είναι πάρα πολύ σε αυτή η περίπτωση ε, που είναι άλλη μια προσέγγιση. Εδώ έχουμε μια γραφική απεικόνηση των χωρικών ορίων και στην περίπτωση της κοφραντίας και της πλυντομή ε, και βλέπετε ότι είναι χωρικά όρια άκρο περιορισμένα, ε, περιορίζονται στην περιοχή όπου λειτουργεί η κοφραντίας και ε, συμμετέχοντες είναι πολλοί στην Κοφραντίας. Όσον αφορά τα χωρικά, τα καινούργια χωρικά όρια, από το 1995, όσον αφορά ε, την διαχείριση των οστράκων από τις 12 από το 1995 καθορίστηκαν τα νέα όρια όσον αφορά τους εταιρισμούς διαχείρισης των στρακών των στεδιών. Λοιπόν, 800 σκάφη έχουν δικαιώματα στην Αδριατική όσον αφορά αυτά το στρακοειδή και υπάρχει κατανομή σε όλη την Αδριατική. Αλλά κάθε ε, συνεταιρισμός έχει συγκεκριμένο χώρο θαλάσσιο ε, που είναι περιορισμένος. Στην περίπτωση τη Κοντζέπα, αναλόγως, έχουμε περιοχές όπου η μέση διάσταση, η παράκτια διάσταση, είναι περίπου 50 ε, χιλιόμετρα κάποιες, συνολικά 500 χιλιόμετρα. Λοιπόν, για τη διαχείριση των στρακοειδών, όσον αφορά τα όρια τα χωρικά, αυτό είναι κάτι που αποφασίστηκε ε, με, σε περιορισμό σε θαλάσσιο χώρο. Τοπικό θαλάσσιο χώρο και αυτοί που έχουν άδεια να αλλιεύσουν τα οστρακοειδή μπορούν να συμμετάσχουν στο consortium ε, και μπορούν να αποφασίσουν τους κανόνες διαχείρισης των αλλιευμάτων. Μόνο όμως αν το 75% ε, των δικαιωμάτων είναι μέσα στο consortium διαφορετικά ε, δεν μπορεί να ισχύσει αυτό το consortium. Χρειάζεται νέα δομή διαχειριστική όλα τα σκάφη, σχεδόν όλα τα σκάφη έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε ένα κονσόρσιουμ. Στην περίπτωση της Κοντζέπα, δηλαδή για τη βιοτεχνική αλεία, είναι άκρως ενδιαφέρουσα η κατάσταση. Διότι δεν προέρχεται από κάποια διάταξη, αλλά αυτή η διαδικασία προέρχεται από ένα άρθρο του Ταμείου Αλίας. Το άρθρο 37 μη προβλέπει τη δυνατότητα διαχειριστικών σχεδίων που θεσπίζονται τοπικά από πλευράς ε, των συνεταιρισμών των αλλίων. Όλα αυτά γίνονται μέσω διαγωνισμού, ανάθεσης και για να, να λειτουργούν αυτά τα consortium πρέπει να περιέχουν 70% των καταχωρημένων αλλιέων σε περιορισμένο συγκεκριμένο χώρο που επιλέγουν οι αλλοίες. Το σχέδιο τοπικής διαχείρισης βασίζεται επί της έρευνας, υποστήριξης έρευνας και της βιολογικής και της οικονομικής και της οικολογικής. Όσον αφορά λοιπόν το δεύτερο σημείο, δηλαδή το δικαίωμα να καθορίζει κανείς, να συντάσσει και να εφαρμόζει κανόνες, όλα τα παρατεθέντα παραδείγματα κατά κάποιο τρόπο μπορούν να καθορίσουν ε, τους κανόνες τους οι κανόνες ουσιαστικά είναι ανάλογοι και θα πρέπει οι κανόνες να είναι λιγότερο περιοριστικοί καινούργια από τους υφιστάμενους και να καθορίζονται οι κανόνες συγκεκριμένα για συγκεκριμένο χώρο αλίας. Θα πρέπει ε, να είναι βιώσιμο το επίπεδο της εκμετάλλευσης που απορρέει από τους κανόνες και να υπάρχει και ανάκτηση των αποθεμάτων, να μειώνονται τα συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων συστημάτων και θα πρέπει να ισχύουν έργα όμνες ένα κανόνες, ο οποίο δεν ισχύει στην πράξη δεν έχει πολύ νόημα. Αυτό ε, είναι κάτι που δεν λαμβάνεται επαρκώ υπόψη, αλλά για να υλοποιηθεί όλα τα παραδείγματα τα οποία εξετάζονται ε, έχουν κάποια προβλήματα. Στην περίπτωση κατά την οποία στην Κοφραντία και την Προυντομή αληθεύει ότι μπορεί να προτείνουν προδιαγραφές στους χώρους αρμοδιότητας κάθε και τη κοφραντία και τη προντομή, αλλά εκ των πραγμάτων αυτό δεν συμβαίνει. Στη Γαλλία συγκεκριμένα για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει οι προδιαγραφές να επικυρώνονται από την αρμόδια νομαρχία. Και αυτό δεν συμβαίνει ποτέ, διότι εφαρμόζεται η διάταξη μια περιορισμένης νομικής ισχύω εφαρμοστικής. Και αν δεν γίνει σεβαστή η διάταξη δεν επιβάλλεται καμία ακύρωση από πλευρά των αρχών. Αντιθέτως, στην περίπτωση το κοσόσιουμ για την ε, βιοτεχνική αλληλεία, όταν το 70% των δικαιούχων αλλιέων μπορούν να συμμετάσχουν στο χώρο, και εκεί δίθεται πρόβλημα της, ισχύω του κανόνος για το υπόλοιπο 30% πέραν από αυτούς που θέλουν να αλλιεύσουν συγκεκριμένο χώρο, διότι σε αυτόν τον χώρο δεν υπάρχει όριο πρόσβασης. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί οι κανόνες που καθορίζονται σε επίπεδο διαχειριστικού σχεδίου τοπικού από πλευράς κάθε κοινότητας αλλιέων θα πρέπει να συμμορφώνεται σε εθνικές διατάξεις. Για να γίνει αυτό ε, θα πρέπει να εγκριθεί η πρόταση για τη διάταξη από τον ίδιο τον Υπουργό και αυτό έχει γίνει τουλάχιστον στην περίπτωση των, της Σικελίας. Όσον αφορά το τρίτο σημείο που χαρακτηρίζει ένα ΤΑΡΦ, το χαρακτηρίζει ποια είναι η συμμετοχή στο ΤΑΡΦ. Στην περίπτωση της Πλουντομή και της Κοφραντίας, η αλληλεία επιτρέπεται μόνο υπό όρους συγκεκριμένους, δηλαδή ο αλληλείας πρέπει να είναι μέλος του ομίλου, αλλά δεν ισχύει όμως τα άλλα δύο κονσόρσιο της διαχείρισης των οστρακοειδών και του κονσόρτσιουμ για τη βιοτεχνική ελεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στην περίπτωση των στεδιών, των μηδιών, χρειάζεται ειδική άδεια. Και μόνο εκείνοι που δεν θέλουν να γίνουν μέλη μπορούν να το κάνουν. Δεν είναι υποχρεωτικό. Εθελοντικά μπορούν να συμμετάσχουν. Όμως εντός του συστήματος διαχειριστικού υπάρχουν κανόνες που προωθούν, δίνουν κίνητρα για τη συμμετοχή στο consortium. Όμως στην πράξη είναι πολύ ε, λίγοι φορείς που παρόλο που έχουν άδεια για την αλληλεία των αεροστακοειδών δεν συμμετέχουν στο consortium. Αυτό για διάφορους ε, λόγους ε, που οδηγούν στο να μην έχει κανείς κίνητρο να είναι εκτός του consortium. Όσον αφορά τη βιοτεχνική αλληλεία όμως, αυτοί που είναι μέλη και είναι καταχωρημένοι στην περιορισμένη περιοχή αλίας ε, συμμετέχουν εθελοντικά. Αν υπάρχουν διαφορές. Όσον αφορά την προάσπιση των δικαιωμάτων, στην περίπτωση της κοφραντίας, επιβάλλονται άμεσα κυρώσεις για όποιον παραβιάσει τους κανόνες και αυτό γίνεται μέσω διαχείρισης της πώληση του προϊόντος στις αγορές όπου γίνεται εκεί διαχείριση αυτών από την κοφραντία. Είναι απλούστατο δηλαδή. Αν τυχαία κάποιο τη κοφραντία αλίευσε ε, παράνομα επιβάλλεται τα μέσα κύριο. Στην περίπτωση της προντομή ε, υπάρχει πολύ μεγάλη νομική ισχύ και έλεγχος. Οι προντομοί δημιουργούνται ε, για να έχουν νομική ισχύ και έλεγχο όσον αφορά την αλία αυτή η εξουσία είναι πολύ αποδυναμωμένη διότι δεν εφαρμόζεται στην πράξη, όμως θεωρητικά θα μπορούσε να υπάρξει αυτός ο έλεγχος και επιβολή των μέτρων. Στην περίπτωση το, της αλίας των οστακοειδών, το κονσόρτσιο μέχρι τη δυνατότητα να ελέγχει και να βάλει κυρώσεις μέσω ε, οικονομικών ποινών τα μέλη μέσω διαδικασία που καθορίζεται και είναι κοινή για όλου τους συμμετέχοντες σε αυτό το κονσόρτσιουμ. Στην περίπτωση όμω για την ε, βιοτεχνική αλία, ε, εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα ε, Τίθεται νόμο, δημιουργείται, θεσπίζεται κρατικό νόμο. Και είναι υπό τον έλεγχο της ακτοφυλακής η αλία. Όσον αφορά τα κίνητρα, από τη στιγμή που δημιουργείται μια νέα περιοχή, νέο τέρφ, δεν αποκλείεται δυνατότητα να εισαχθεί ένα τέρφ καινούριο στην ε, Μεσόγειο. Από τη στιγμή που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ταιριάζει στη Μεσόγειο, ε, ατομικότητα υπάρχει, ε, υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Και εκεί που δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν φυσιολογικέ ομαδοποίησει, χρειάζεται πίεση, άρα χρειάζεται να δοθούν κίνητρα για να δημιουργηθούν οι ομαδοποίησει. Όσον αφορά ε, συμπράξεις ε, για, για τα στοακοειδή υπάρχουν ε, μέτρα διαχείριση για να ξεκινήσουν αυτές οι συμπράξεις και θα πρέπει ε, αντί να εισαχθούν κανόνες για τη μείωση του δυναμικού παρόλο που είναι σημαντικοί κανόνες οι οικονομικοί πόροι περισσότερο κατευθύνονται παρόλα αυτά στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του διαχειριστικού οργανισμού, διότι χωρίς αυτή την αξιοπιστία προφανώς είναι δυσκολότατο να μπορεί να λειτουργήσει μια περιοχή αλίας, ένα turf. Ε, όσον αφορά όμως ε, άλλους φορείς αναλόγως υπάρχει λύση διαφορετική. Αλία πιο ανοιχτή στα Χρειάζεται διαχείριση κάθε συνεταιρισμού, κάθε consortium μέσω ορίων που θεσπίζονται, στόχοι τίθενται για την αποκατάσταση των αλλιευμάτων και καθορίζονται αναγκαίες δράσεις για να αρθούν τα όρια όταν δεν χρειάζονται. Αυτά περιέχονται στο πραγματισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας. Και οι κοτζέπα αυτοί έχουν προτεραιότητα όσον αφορά την ενεργοποίηση των διαγωνισμών ανάθεσης για να εφαρμόσουν τα διάφορα προγράμματα που από το Ταμείο Αλίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι είναι συγκεκριμένο κίνητρο που δίνεται για να ομαδοποιήσει, να συμμετέχουν οι αλλοί σε τέτοιους φορείς. Όλο αυτό το πρώτο τμήμα που πράγματι είναι μακρό, αυτή η εισαγωγή χρησιμεύσε για να δείτε ποια σχέση υπάρχει μεταξύ πολιτική αυτών των χώρων αλληλεία του ΤΕΡΦ με την κοινή αλληλευτική πολιτική. Ένα ΤΕΡΦ, λοιπόν, ένα ΤΕΡΦ εξαλείφει την ανάγκη μικροδιαχείριση σε επίπεδο κοινοτικό. Αυξάνει και τις ευθύνες των αλλιέων, των εμπορευομένων, προς όφελος μιας προσέγγισης με στόχο το τελικό αποτέλεσμα και αυτά είναι χαρακτηριστικά που διαπιστώσαμε να υπάρχουν κατά την εφαρμογή των TERF για ε, βιοτεχνική αλληλεία. Μπορεί να υπάρχει διαφοροποιημένο καθεστώς που εφαρμόζεται, υπάρχουν διαφοροποιημένα καθεστώτα. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν κομμάτι ε, των προτάσεων της νέας αλληλευτικής πολιτικής που ήδη έχουν ενσωματωθεί στις δραστηριότητες τις οποίες προανέφερα. Πρώτο συμπέρασμα από όλα αυτά. Ένα ΤΕΡΦ, μια περιοχή αλεία, μπορεί να είναι ένα εργαλείο πολύ ενδιαφέρον στην περίπτωση της μικρή κλίμακα παράκτη αλεία, Δεν υπάρχει μια και μοναδική συνταγή, μια μοναδική λύση. Πρέπει τα ΤΕΡΦ να οριοποιούνται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και ένα τάρφ δεν μπορεί να εισάγεται πάντα καινούριο. Σε πολλέ περιπτώσει είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι αποτελεσματικό κάτι τέτοιο. Δεν πληρούνται οι προποθέσει για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο χώρο, ένα τερφ. Δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτό το μέτρο. Και τέλο, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι παρά το άρθρο 37M του Ταμείου Αλίας προτείνει αυτό το τρόπο διαχείριση τοπικό επίπεδο, δεν υπάρχει ε, ουσιαστικά ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, regulatory framework, κάποια διάταξη νομοθεσία που να καθορίζει λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας. Και αυτό είναι ένα όριο ε, που θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε στο μέλλον, ελπίζω. Όσον αφορά τη Μεσόγειο, ερχόμαστε τώρα στη Μεσόγειο, στα μεσογειακά θέματα. Φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε το 1980, από την πρώτη έκθεση της ΦΑΟ, ε, και μετά με άλλη έκθεση η Επιτροπή την Αλία στη Μεσόγειο πάντα υποστήριζε την ανάγκη διαχείρισης της αλίας στη Μεσόγειο μέσω της αληθικής προσπαθίας. Δηλαδή δυναμικό αλίας, στόλος, δραστηριότητα, χρόνος αλίας. Ε, και αυτό ίσχυε επί πολλά χρόνια, αλλά είδαμε ότι αυτή η προσέγγιση δεν έδινε πάντα ικανοποιητικούς καρπούς και διότι στην περίπτωση πολλαπλών ιδιαιτεροτήτων δεν υπήρχε συσχετισμό μεταξύ ε, αφοπλισμού σκαφών, παροπλισμού σκαφών, όταν θέλαμε να μειώσουμε το δυναμικό, δεν υπήρχε συσχετισμό με την αλευτική προσπάθεια, διότι υπήρχαν πολλές ιδιαιτερότητε και ίδιοι και μπορούσαν να έχουν το ίδιο αλίευμα διαφορετική τρόποι αλλίες. Οπότε δεν ήταν εύκολο να προσαρμοστεί, στοχευμέ, να, να εφαρμοστεί στοχευμένη πολιτική. Και χρονικά είναι δύσκολο, να διαχειριστεί κανείς την επόμενη περίοδο και ο γόνος να διαφυλαχθεί. Σημειώνεται ότι η τεχνολογική πρόοδος ε, ε, τίνει να αυξήσει την προσπάθεια, οπότε η συνεχής μείωση του... Έχουμε μείωση του δυναμικού και από την άλλη βελτίωση τεχνολογία που αυξάνει την προσπάθεια. Άρα η μείωση του δυναμικού δεν οδηγεί απαραίτητα σε μια ικανοποιητική πολιτική όσον αφορά τη διαφύλαξη των πόρων. Όσον αφορά το Μεσόγειο, το πιο ενδιαφέρον τμήμα συνδέεται με την τροποποίηση της όλης πολιτικής. Ο κανονισμός για τη Μεσόγειο 1967-06 ε, προτείνει τρία συγκεκριμένα στοιχεία. Τεχνικά μέτρα, εθνικά σχέδια διαχείρισης και κοινοτικά σχέδια διαχείρισης. Είναι τρία στοιχεία που διαφέρουν το ένα με το άλλο και απαιτούν ε, προσοχή. Όσον αφορά τα εθνικά σχέδια. Η Ιταλία έχει συλλέξει κάποια εμπειρία, αποκομίσει κάποια εμπειρία. Ήταν ανάμεσα στις λίγες χώρες που παρουσίασαν διαθρωμένα σχέδια. Σύμφωνα με τη διάταξη και η προσέγγιση που ακολουθήθηκε ήταν τυπική, standard. Παρήχθησαν οκτώ σχέδια για την αλία με, με ε, σχέδια διαχείρισης με το παραγάδι και στη δίβλο της Σικελίας με διάφορα είδη. Με, με και δράγες. Λοιπόν, όλα αυτά εξελίσσονται διότι κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητες και οι τρόποι αλλιές προσαρμόζονται. Τα σχέδια για να ανταποκρίνονται σε εθνικό επίπεδο ε, θα πρέπει να βασίζονται σε γεωγραφική υποδιέρεση GSA της ΦΑΟ. Ε, δεν υπάρχει ομοιογένεια μεταξύ των διαφόρων χώρων. Ε, οι δείκτε ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή. Άρα αυτό μα οδηγεί σε διαφορετικέ διαδικασίε που πρέπει να ακολουθούν για καλυφθεί κάθε περιοχή. Εδράζονται επί κατά προσπάθεια ε, και κάθε σχέδιο λοιπόν εμπεριέχει ένα κομμάτι που αφορά την ε, οριστική πάυση, ε, μέτρα όσον αφορά το μάτι των δικτύων κλπ, ε, χώρους για την ανάπτυξη γόνου κλπ. Υπάρχουν πολλαπλά σχέδια, που, πολλαπλά μέτρα σε κάθε σχέδιο. Κίνητρο τώρα για προσέγγιση κατά υποπεριοχές εδράζεται επί ασυνήθιστο για τη Μεσόγειο, κάτι ασυνήθιστο για τη Μεσόγειο, ευασίζεται η προσέγγιση σε πολλά στοιχεία, πολλές πληροφορίες μετά από τον κανονισμό για τη συλλογή στοιχείων. Αλλά πριν το data collection, ε, πριν τους κανονισμούς για τη συλλογή ε, στοιχείων υπήρχαν πάρα πολλές πληροφορίες. Και καμιά φορά τα στοιχεία που δημοσιεύονται όμως δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα που επικρατεί στη Μεσόγειο. Η κατανομή κατά GSA ε, ε, εξαρτάται από ιδιαιτερότητε. και μπορούν να δοθούν οικονομικοί πόροι σε κάθε GSA μέσω εθνικού προγράμματος αν γινόταν αυτό σε εθνικό επίπεδο η κατανομή των πόρων δεν θα γινόταν με αποτελεσματικό τρόπο. Εδώ μπορείτε να δείτε γιατί κάναμε την επιλογή. Λοιπόν, τι γίνεται στην περίπτωση ε, του μπαρμπουνιού και της κόκκινης γαρίδας βλέπετε στην Αδριατική πώς γίνεται χωρίς. Στο κάτω, στην κάτω Αδριατική, στην νότια Αδριατική έχετε τάσεις που είναι διαφορετικές που αλλάζουν συνεχώς. Όσον αφορά όμως το τυρινικό πέλαγος, σε σύγκριση με την Σικελία, τη Βόρεια, ε, και εκεί στην περίπτωση της Γαρίδας από 200-800 μέτρα βάθος πάμε για την Ελία. Ε, και βλέπετε ότι υπάρχουν διαφοροποίησεις. Άρα ε, χρειάζονται ειδικά μέτρα για να καλυφθεί αυτό. Στην περιοχή των οικονο... στον τομέα οικονομικών παραμέτρων, ε, όγκος εκφορτώσεων, σε διαφορετικές περιοχές με το ίδιο σύστημα, ε, βλέπετε ότι υπάρχουν διαφορετικές ε, συμπεριφορές. Αλλά σχετίζεται και με το απόθεμα και στην ίδια υποπεριοχή βλέπετε συμπεριφορές μικρής κλίμακας σε πιο μεγάλη αλία βλέπετε ότι υπάρχουν διαφοροποίησεις που οφείλονται και στις τιμές, σε αλλαγές στις τιμές και στις μεγάλες διακυμάνσεις που υπάρχουν από χρονιά σε χρονιά που ε, οι διακυμάνσεις καθορίζουν και τις αποφάσεις των αλλιευτικών επιχειρήσεων που βασίζονται επί των τιμών. Είναι αποτελεσματικά λοιπόν τα εθνικά διαχειριστικά σχέδια βάσει της εμπειρίας ε, που έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα. Μιλάμε για σχέδια που εδράζονται επί της προσπαθίας. Άρα ε, περιέχονται τα όρια που προαναφέραμε. Τα όρια της προσπαθίας. Και στα πλαίσια των σχεδίων αυτών το permanent withdrawal και η προσωρινή πάυση και η μόνιμη πάυση ε, είναι σημαντικά εργαλεία παρέμβασης αλλά θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες. Τώρα προσπαθώ να προχωρήσω γρήγορα, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι εύκολο να παρακολουθήσετε πιθανότατα την παρουσίαση, διότι είναι πολύ ευρύ το θέμα τους ε, Μεσογείου. Βλέπετε, στο ενώ της Σικελίας είχαμε ενδιαφέροντα αποτελέσματα όσον αφορά την οριστική πάυση. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι είναι στο ίμιση η αλία τελευταία δέκα χρόνια. Μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού της οριστικής παύσης έχουμε μία μείωση του δυναμικού σε σχέση με τον στόχο που είχε το διχειστικό σχέδιο. Προβλεπόταν μείωση 25% της ελευτικής προσπάθειας όσον αφορά το δυναμικό αφορά τη γαρίδα. αυτός ο στόχος και τα ωφέλη εντοπίστηκαν, εντοπίστηκαν στην περίπτωση της αλίας λοιπόν της γαρίδας σε μεγάλο βάθος είδαμε αύξηση ε, του αποθέματος. Ταυτόχρονα όμως είχαμε μία μείωση της αλλιευτικής πίεσης στις παράκτιες περιοχές. Διότι τα σκάφη που αλίευαν παρακτίους μετακινήθηκαν και πήγαν εκεί όπου πετυχαίναν τα αποτελέσματά τους. Άρα ο στόχος επετεύθη. Όμως δυστυχώς εξουδετερώθηκε, διότι πώς να το πω, ήταν ένα όριο που είχε τεθεί που δεν ε, έλαβε υπόψη άλλες όρους. Εφόσον είναι δυνατόν να μετακινηθούν τα σκάφη σε άλλες αλληλευτικές περιοχές, διαφυλάξαμε μεν τη, τη γαρίδα, αλλά όπως βλέπετε, θα το δείτε σε λίγο, η θνησιμότητα η εθνισιμότητα της γαρίδας που είναι στο γαλάζιο αυξήθηκε διότι υπήρξε συγκέντρωση των ε, σκαφών σε αυτή την περίπτωση. Ενώ όσον αφορά ε, το σγόμπρο ε, είχαμε άλλο αποτέλεσμα. Πετύχαμε λοιπόν όσον αφορά τον μπαρμπούνι είχαμε άλλα αποτελέσματα. Λοιπόν, όσον αφορά τα σχέδια τα κοινοτικά της διαχείρισης και τις προδιαγραφές, terms of reference, που αφορούσαν την ανάλυση ε, της αλίας στο GSA 17 βλέπετε και το κοινοτικό σχέδιο που αφορούσε την GSA 17 ε, Μέση Αδριατική με Βόρεια Αδριατική και εκεί η Κροατία μπορεί να, όταν θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί αυτό το διαχειριστικό σχέδιο το οποίο ε, αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες ε, μεγάλη διαφορά που υπάρχει, δηλαδή διαθωτική όσον αφορά την παραγωγή. Στην Κροατία αλλιεύουν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στην Ιταλία. Λοιπόν, αυτό έχει συνέπειες η διαφοροποίηση τρόπου αλλιές όσον αφορά την εφαρμογή ενός διαχειριστικού σχεδίου. Όσον αφορά την πελαγική αλλία. Έχει εγκριθεί πρόσφατα μία μέθοδος για την διατύπωση των σχεδίων διαχείρισης για τη μικρή πελαγική αλία στην Ιταλία και το σχέδιο αυτό είναι ένα modus operandi το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα μπορέσει να γίνει αποδεκτό και από άλλες περιοχές. Είναι εν πάση περιπτώσει ένα πρώτο πείραμα για ένα σχέδιο διαχείρισης που μπορεί καταρχήν πέραν του Ιταλικού στόλου να χρησιμοποιηθεί και από άλλους αλληλευτικούς στόλους. Η ιδιαίτερη δύναμη κατά κάποιο τρόπο της περιοχής της Αδριατικής είναι η δυνατότητα να υπάρξει ένα ενωσιακό σχέδιο αλίας όπως το Αντριαμέντ της ΦΑΟ μέσα στο οποίο μπορεί να τίθεται από κοινού η επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και να υπάρξει και κοινή διαδικασία αξιολόγησης των αλλιευτικών αποθεμάτων. Επομένως, η χρήση αυτών των κοινοτικών σχεδίων διαχείρισης μπορεί να βασίζεται σε κοινού ορισμούς και σε κοινέ μεθόδους αξιολόγησης. Έρχομαι στο δεύτερο και μόνο συμπέρασμα ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια σημαντική βελτίωση της προηγούμενης πολιτικής, η οποία μέχρι στιγμής βασιζόταν μονάχα στον έλεγχο της αλληλευτικής προσπάθειας. Αλλά δεν έχουμε ακόμα φτάσει σε ένα σύστημα το οποίο θα μπορέσει να εφαρμόσει περιορισμούς για τη χρήση αλλιευτικών μεθόδων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, ακόμα και αυτά τα σχέδια διαχείρισης δεν θα ευδοκιμήσουν. Αν όμω είτε η πρόταση Κομισιόν είτε οι τροπολογίε του Κοινοβουλίου εισαγάγουν την έννοια του δικαιώματο χρήση αλλιευτικών μεθόδων, έχουμε μια σημαντική καινοτομία. Και υπάρχει μια σειρά από επιχειρήματα σε σχέση με το σενάριο αυτό του να συνδυάσουμε ένα turf που έχει εδαφική βάση βέβαια με συγκεκριμένες ποσοστώσεις για αλίευση. Θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να είναι ένα εγχείρημα ενδιαφέρον, αλλά παραμένουν πολύ μεγάλες ανισομέρειες και διαφορε... διαφορές από περιοχή σε περιοχή. Νομίζω ότι οι αλληλευτικές κοινότητες οι οποίες ενδιαφέρονται για ένα turf, ένα turf δεν μπορούν να είναι πάντα οι ίδιες οι οποίες θα αναλάβουν τις αποφάσεις σε σχέση με τα πρότυπα τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν και δεν μπορεί το ΤΕΡΦ μόνο και μόνο να καθορίσει την πρόσβαση στους αλληλευτικούς πόρους. Χρειάζεται μια ευρύτερη αντιμετώπιση και αυτό το θέμα θα πρέπει να διαλευκανθεί. Κάτι άλλο όμως το οποίο για μένα είναι σημαντικό είναι το θέμα της μη δυνατότητας μεταφοράς των αλληλευτικών ποσοστώσεων. Αυτό είναι μια θέση που είναι θεμητή βέβαια. Το πρόβλημα το οποίο προκύπτει είναι ότι αν δεν είναι μεταφέρσιμες, μεταφερόμενες οι ποσοστώσεις και χωρίς ένα σχέδιο για τη μείωση των αλλιευτικών στόλων, ένα σύστημα αχρήστευσης αλλιευτικών πλήρων, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτύχουμε τη μείωση της αλλιευτικής ικανότητας, γιατί σε μια αγορά χωρίς συγκέντρωση και χωρίς μεταφορά ε, ποσοστώσεων θα μειωθεί. Δεν θα υπάρχουν οι δυνατότητες αυτές αλίας και δεν θα υπάρξει έτσι η δυνατότητα να μειώσουμε την αλλιευτική ικανότητα. Θα ήθελα λοιπόν, ήθελα απλώς να αναφέρω όλα αυτά τα στοιχεία, τις πτυχές που είναι σημαντικές, αλλά... Η μόνη πτυχή που μπορεί να ενδιαφέρει είναι ότι η ποσόστοση ε, είναι αποτελεσματική στην περίπτωση που σχετιζόμαστε με ένα είδος αποθέματος. Ε, η κοινή ιδιοκτησία και ο συναγωνισμός μεταξύ των σκαφών ε, έτσι αφαιρείται και αφαιρείται και ο αγώνας ε, για την αλία και για τις επενδύσεις. Απ' την άλλη πλευρά, οι παραγωγείς μπορούν να συνδυάσουν αποτελεσματικά τους παραγωγικούς παράγοντες. Δηλαδή, εκεί όπου υπάρχει ένα είδος αποθέματος, η ποσόστος προσπάθειας μπορεί να θεωρηθεί σαν μία λύση χρήσιμη για την καλύτερη διαχείριση. Το ίδιο όμως δεν αληθεύει στην περίπτωση της ποσόστοσης του αλλιεύματος. Της προσπαθία, μάλλον, της τη προσπαθία, Διότι η προσπάθεια λειτουργεί επί του χρόνου αλλία. Δηλαδή, στόχο του αλλιεύματο θα είναι η μονάδα χρονική τη αλλία αυτή η χρονική μονάδα θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί το εισόδημά του. Οπότε παραμένει υψηλή συνιστόσα συναγωνισμού στη δραστηριότητα, συναγωνισμού σε χρονικό επίπεδο. Οπότε δεν επιλύεται το πρόβλημα ε, της αποτελεσματικής διαχείρισης και της απόδοσης. Πιθανότατα λοιπόν η ποσόστοση της προσπαθίας στην περίπτωση πολλαπλών ειδών είναι το καλύτερο πλέον δεδειγμένο εργαλείο, αλλά θα πρέπει να συνδέεται με άλλε διαχειριστικέ ρυθμίσει, όπω το να διαμορφώνονται οι μέρε αλληλεία, οι ώρε τη αλληλεία, συναρτήσει τη αυθονία του αποθέματο. Διότι μόνο ότι ο τρόπο είναι δυνατόν να γίνει μια αποτελεσματική διαχείριση. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη αν πήρα λίγο χρόνο παραπάνω. Στα συμπεράσματα μπορούμε να πούμε ότι αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε όσον αφορά τη μικρή κλίμακα αλληλεία μπορούμε να παρέμβουμε πάνω απ' όλα μέσω του δικαιώματος χρήσης εδαφικού ευχόμενοι ότι μπορεί να υπάρχει τυπική διαφοροποίηση να υπάρχει μια διαδικασία για τα τοπικά διαχειριστικά σχέδια και να, τα TERF μαζί με τοπική διαχείριση να είναι ενδεχομένω μια λύση στην περίπτωση της κλίμακα, μικρής κλίμακας αλίας, στην περίπτωση μη κοινών αποθεμάτων όπου εκεί ε, επηρεάζει εδαφικός διαχωρισμός, εκεί θα ήταν δυνατόν να εισαχθεί ένα turf υπό τον όρο όμως ότι οι κανόνες αποφασίζονται από τους ίδιους τους αλείς, αλλά αυτό πιστεύω ότι ε, δύσκολα μπορεί να ισχύσει. Λοιπόν, τι επομένει. Τα διαχειριστικά σχέδια τεχνικά όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 19 του κανονισμού του κοινοτικού για τη Μεσόγειο, ίσως είναι το πλέον δεδειγμένο μέτρο. Στην περίπτωση όμως των κοινών αποθεμάτων, των κοινών στόκ, εκεί τα εδαφικά όρια, τα χωρικά όρια ε, έχουν κάποια επιρροή και συνεπώς δεν είναι δυνατό να μην ληφθούν υπόψη. Είδαμε μια περίπτωση του Community Level Management Plan που προβλέπει το άρθρο 18 για τον κανονισμό ε, του GSA 17 δηλαδή όπου εκεί υπάρχουν κοινοτικά κράτη όπως και όταν μπει η Κροατία ε, μπει στην Ένωση θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τέτοιου είδους προσέγγιση και δραστηριότητα προφανώς στην περίπτωση των αποθεμάτων σε διεθνείς χώρους παρόλο που αυτό δεν είναι ακόμα δεν συμπεριλαμβάνει τι προδιαγραφέ που έχουν καθοριστεί. Αληθεύει σε διεθνή ύδατα ισχύει η αλληλεία ενό μοναδικού είδου κάθε φορά. Άρα εκεί χρειάζεται διαχείριση μέσω ποσοστώσεων αλλιευμάτων που θα μπορούσαν να θεσπιστεί. Αυτό είναι μια διαστηριότητα που θα αφορά περισσότερο το GRCM. Συνοψίζοντας λοιπόν, στην περίπτωση των μη κοινών αλλιευμάτων, στις, στην παράκτη αλληλεία ε, έχουμε το τα βασικά εργαλεία που είναι τα εθνικά σχέδια τα αλλιευτικά, National Fisheries ε, Plans, χρειάζεται να υπάρχουν ε, εθνικά αλλιευτικά δικαιώματα. Με τα πελαγικά είδη όμω υπάρχει διαφοροποίηση μέσω α, ποσοστώσεων προσπαθίας και αλληλεία. Αυτά δεν μπαίνουν όμως στη δυνατότητα μεταφορά σε αυτή την περιπτώση. Αναφέρομαι στην τροποποίηση του Κοινοβουλίου εδώ. Στην περίπτωση της αλίας πελαγικών ειδών, ποσοστός προσπαθίας και ποσοστώσεις αλίας. Στην περίπτωση όμως των ε, ε, ε, ειδών που ζουν σε βάθος, ε, εκεί η διαχείριση μπορεί να γίνει ε, μέσω ποσοστώσεων προσπαθίας με διορθώσεις που προανέφερα. Δηλαδή με αυτόματα εργαλεία καθορισμού ημερών αλίας συναρτήσει δικτών ε, προστασίας της βιομάζας από τον ένα χρόνο στον άλλον, των αποθεμάτων δηλαδή. Στην περίπτωση των κοινών αποθεμάτων, των κοινών αλληλευμάτων, εξαφανίζονται τα τόρφ αλλά δεν διαφοροποιείται ο τρόπος διαχείριση. Όταν μιλάμε υπελεγγυκά, ήδη βάζουν δεν βάζουν ποσοστώσεις προσπαθίας και αλλιευμάτων. Καθορίζουμε το χρόνο αλίας και ταυτόχρονα την ποσότητα του αλλιεύματο. Στην περίπτωση των ειδών μεγάλου βάθους, πιο αποτελεσματικό μέσο θα έπρεπε να είναι αυτό που εδράζεται επί των ποσοστώσεων προσπαθίας, ε, προσπαθίας ξεχωριστών για κάθε είδους. Συγγνώμη που μίλησα πολύ γρήγορα, μου βάλατε, μου αναθέσατε ένα έργο τεράστιο, οπότε υπήρχε κάποιο πρόβλημα να μπορέσω να συνοψίσω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σπανιόλο. Όντω, μακρηγορήσατε, αλλά με ιδιαίτερη χαρά παρακολουθήσαμε την παρουσίασή σα. Περνάμε τώρα στον επόμενο εισηγητή μα, επόμενο καλεσμένο μα, που είναι ο Χουαν Λουί Σουάρε Δεβιβέρο. Ε, θα του δώσω το λόγο χωρί άλλη καθυστέρηση, αλλά το θέλουμε παρακαλώ να μην μακρηγορήσει όπω ο πρώτο μα εμπειρογνώμονα, γιατί δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο στη διάθεσή μα. Παρακαλούμε, κύριε Σουάρε Δεβιβέρο. Profesor, tiene Έχετε το λόγο κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ και καλημέρα σας. Η δική μου παρουσίαση αφορά την διεθνή συνεργασία και ιδιαίτερα τη συνεργασία στη Μεσόγειο σε σχέση με τις αλληλευτικές δραστηριότητες. Αν υπάρχει ένας όρος ε, που προσδιορίζει και χαρακτηρίζει καλύτερα συνοπτικά την ε, Μεσογειακή Λεκάνη είναι η περιπλοκότητα. Πολιτική, δικαιοδοτική και κοινωνικο-οικονομική περιπλοκότητα. Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα στα θέματα συνεργασίας και διεθνών σχέσεων. Ως ε, οι λεκάνες υδάτινες, ε, η Μαύρη Θάλασσα και η Μεσόγειος ε, αντιπροσωπεύουν μόνο το 1% η Μεσόγειος για παράδειγμα των ωκεανών αλλά παρά την ε, περιορισμένη έκθεσή τους οι δύο λεκάνες στις δύο αυτές λεκάνες συναντιόνται τρεις Ήπειροι η Αφρική, η Ασία και η Ευρώπη Κάτι που δημιουργεί πολλές φορές μεγάλες εντάσεις. Ένα είδους ε, γεωγραφικού στρες δηλαδή, όπως λέμε. Κάτι που εξηγεί και την περιπλοκότητα και τις δυσκολίες διαχείρισης των ε, κοινών πτυχών των δύο αυτών ε, υδάτινων λεκανών, της Μεσογείου και του Ευξηνού Πόντου. Ένα από τα αποφασιστικά στοιχεία της συνεργασίας και για τις δύο αυτές λεκάνες και ιδιαίτερα όμως για τη Μεσογειακή λεκάνη είναι αυτό το κοινωνικο-οικονομικό χάσμα όπως λέμε που υπάρχει μεταξύ της βόρειας και της νότιας όχθης της Μεσογείου. Στην περίπτωση αυτή, στη Μεσόγειο, η σχέση αυτή είναι ένα προς 23,5%. 1 προς 23,5 συγγνώμη. Και τα βασικά άκρα είναι η Γαλλία και η Αίγυπτος. Η Γαλλία είναι η πιο πλούσια χώρα, ενώ η Αίγυπτος είναι η χώρα με τα λιγότερα, λιγότερα εύπορη χώρα στη Μεσόγειο. Ενώ στην, στη Μαύρη Θάλασσα έχουμε μεγαλύτερη ομοιογένεια. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλο κοινωνικό-οικονομικό χάσμα. Είναι 1 προς 4,7. Έτσι εξηγούνται σε κάποιο βαθμό οι δυσκολίες της κοινή διαχείρισης και οι δυσκολίες στη συνεργασία και στις δύο αυτές ειδωτινές λεκάνες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία για τα αλληλευτικά θέματα. Συνεργασία στην αλληλεία. Ένα από τα κέρια σημεία είναι η δικαιοδοτική διάρθρωση του ευξήνου πόντου και της Μεσογείου αφετέρου. Και ίσως το πιο αξιοσημείωτο εδώ θέμα, στη Μεσόγειο ειδικά, είναι η ποιοτική και ποσοτική αλλαγή που διαπιστώθηκε τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα θα λέγαμε η αλλαγή που έχει συντελεστεί τους τελευταίους μήνες λόγω της σταδιακής δήλωσης των αποκλειστικών δικαιωμάτων. Αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τη Μεσόγειο που μέσα σε λίγο καιρό, μέσα σε λίγους μήνες ουσιαστικά, περάσαμε από, την ανοιχτή θάλασσα που ε, κυριαρχούσε το 40% των νερών, μειώθηκε σε ένα 30% λόγω της ε, διακήρυξης των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Επιπλέον όμως ε, στη Μεσόγειο έχουμε και μεγάλη πολυμορφία των ε, νομικών καθεστώτων. Πέραν των ε, αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, έχουμε ζώνες ε, προστασίας αλίας και ζώνες οικολογικής προστασίας. Στην περίπτωση της Μαύρης Θάλασσας, όλη η την που είναι σχετικά περιορισμένη, υπόκειται στη δικαιοδοσία των παράκτιων χωρών. Θα ήθελα επίσης να τονίσω το βάρος που φέρει στη διαχείριση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το, ποσό, το, ποσοστό των υδάτων που εμπίπτει στην εθνική δικαιοδοσία είναι της έξω του 34%. Υπάρχει περιθώριο αύξησης. Μια και αναμένεται η ένταξη της Κροατίας ως ονούπο αλλά και ε, η Ιταλία μπορεί να διευρύνει τα χωρικά της ύδατα, όπως και η Ελλάδα. Εκεί όμως είναι πιο δύσκολο λόγω της ε, αντιδικές που υπάρχει με την Τουρκία. Πάντως, ε, πολύ σύντομα, το δικαιοδοτικό βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Μεσόγειο θα υπερβαίνει το 40% των υδάτων της Μεσογείου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί δίνει έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές δυνατότητες και περιθώριο δράσης στη Μεσογειακή Λεκάνη. Στην Μαύρη Θάλασσα το δικαιοδοτικό ποσοστό, η δικαιοδοτική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ μικρότερη, είναι της τάξης του 14%. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατάσταση αλίας ε, σε ένα κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Μεσόγειος δεν ε, έχει ιδιαίτερο βάρος ό,τι αφορά την ανάπτυξη της βιομηχανικής αλίας. Σε σχετικούς όρους βέβαια διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο και είναι μια πηγή εσόδων ε, για τις τοπικές και περιφερειακές κοινότητες. Και φυσικά έχει ιδιαίτερη ζήτηση ε, στον τουρισμό η περιοχή αυτή. Εδώ έχουμε τρία βασικά χαρακτηριστικά της αλληλείας στη Μεσόγειο που μας δίνουν μια ισορροπία σε ό,τι αφορά τα αλλιεύματα τα αλλιεύματα του Ευρωπαϊκού Ελευτικού Στόλου και τα αλλιεύματα των στόλων των άλλων παράκτων χωρών της Μεσογείου. Σε ό,τι αφορά την εδαφική παρουσία, έχουμε μεγαλύτερη παρουσία των χωρών του Νότου και της Ανατολής, αλλά σε ό,τι αφορά την κατανάλωση των αλλιευτικών προϊόντων, διαπιστώνουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κατανάλωση είναι πολύ μεγαλύτερη. Κάτι που ε, δείχνει την μεγαλύτερη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και από τους αλληλευτικούς πόρους αλλά και από τις εισαγωγές σε αλληλευτικά προϊόντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατάσταση της διεθνούς συνεργασίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια κατάλληλη νομικοθεσμική δομή Έχουμε πάνω από 60 διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες και έχουμε και ένα ολόκληρο δίκτυο φορέων ε, και οργανισμών που καταρχήν θα μπορούσαν να εγγυηθούν μία αγαστή συνεργασία. Παρ' όλα αυτά, όλο αυτό το νομικοθεσμικό οικοδόμημα, όλη αυτή η διάρθρωση νομικοθεσμική δεν εξασφαλίζει μία αποδεκτή οικολογική κατάσταση γιατί ιδιαίτερα στη Μεσογειακή Λεκάνη έχουμε μια πολύ χαλαρή πολιτική ολοκλήρωση. Επίσης διαπιστώνουμε αισθητές διαφορές μεταξύ Βορρά και Νότου. Στο Βορρά έχουμε πολύ μεγαλύτερη οργάνωση και ολοκλήρωση χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στη Νότια Όχθη πολύ λιγότερη ο συντονισμό και συνεργασία. Κάτι που δυσχεραίνει την συλλήψη αποφάσεων και, της, και τη διαμόρφωση συνένεσης για τη διαχείριση θεμάτων της Μεσογείου που είναι κοινού ενδιαφέροντος. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ε, το αυξανόμενο βάρος των κοινοτικών θεσμικών οργάνων στις περιφερειακές θάλασσες. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπο λειτουργία των διεθνών σχέσεων μας οδηγεί στην εφαρμογή και την εκτέλεση των αδειών ε, να εμπίπτουν σε κάθε κράτος. Κάτι που δημιουργεί ένα μεγάλο κατακαιρματισμό ε, στην Μεσόγειο ειδικά, γιατί είναι πολλές ε, οι χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο. Είχαμε πρόσφατα πολλές μελέτες ε, που έγιναν μετά από έτοιμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που όλες ζητούν τη δημιουργία ενός φόρουμ για να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων. Τώρα, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της έρευνας στην Αλία στη Μεσόγειο που ήταν ένα από τα θέματα και μία από τις ερωτήσεις στο σημείο μας για την παρουσίασή μου. Νομίζω ότι τα εργαλεία που επιτρέπουν την ανάπτυξη της έρευνας ε, για την Αλία στη Μεσόγειο και οι μηχανισμοί αυτοί είναι προσωρινού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη πιο μακροπρόθεσμων και μακρόπνων ερευνητικών σχεδίων και προγραμμάτων. Άλλωστε, δεν υπάρχει και μία χρηματοδοτική δομή που να εξασφαλίζει μία σταθερότητα στην ανάπτυξη των ερευνητικών σχεδίων για την αλία. Επιπλέον, με την σοβούσα οικονομική κρίση το θέμα χερίνει ακόμη περισσότερο και επιτείνεται αυτή η αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά του εθνικού προπολογισμού. Γιατί οι εθνικοί προπολογισμοί χρηματοδοτούν αυτά τα ερευνητικά σχέδια για την Αλία. Οπότε εδώ βλέπουμε πως και στις δύο λεκάνες, και στη Μεσόγειο και στην Μαύρη Θάλασσα, έχουμε πλήρη κάλυψη από αυτά τα προγράμματα έρευνα για την αλία, που χρηματοδοτούνται όμω η τελική ανάλυση μόνο από τρει χώρε. Σε συνεργασία φυσικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε το τελικό αποτέλεσμα οδηγεί σε μια μεγάλη εξάρτηση της έρευνας από ένα μικρό αριθμό χωρών και φυσικά από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Από αυτά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η επιβίωση των προγραμμάτων αυτών. Ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της έκθεσης είναι να κρίνουμε ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση στην αλληλευτική συνεργασία, η διμερής ή η περιφερειακή. Θα μπορούσαμε ίσως να βρούμε την απάντηση στην ερώτηση αυτή απαντώντας προηγουμένως σε τρεις ερωτήσεις για τους πόρους, τις δικαιοδοσίες και την εθνική δράση. Σε ό,τι αφορά τους πόρους, θα έπρεπε να διαπιστώσουμε ότι ένα μεγάλο τμήμα των αλληλευτικών πόρων στη Μεσόγειο είναι κοινή πόρη, κοινή αλληλευτική πόρη. Κάτι που προϋποθέτει φυσικά μια περιφερειακή προσέγγιση και εστίαση. Αναλύοντας τις τάσεις σε ό,τι αφορά την διαχείριση βλέπουμε ότι μία από τις προτάσεις ε, που εξετάζονται τα τελευταία χρόνια είναι η κατάταξη και οργάνωση με βάση τα οικοσυστήματα. Αυτή η κατάταξη με βάση τα οικοσυστήματα και η οργάνωση με βάση τα οικοσυστήματα προϋποθέτει επίσης μία περιφερειακή ή υποπεριφερειακή προσέγγιση και συνεργασία. Σε ό,τι αφορά τώρα τις δικαιοδοσίες, Έχουμε μία τάση για εθνικοποίηση των χωρικών υδάτων. Κάτι που ευνοεί περισσότερο τη σύναψη διμερών συμφωνιών. Ενισχύεται δηλαδή εδώ η διμερής προσέγγιση σε σχέση με την περιφερειακή. Τώρα, αν ανακύπτει το ερώτημα διανύει η κρίση η περιφερειακή δράση δεν υπάρχουν αποδείξεις στην ειδική βιβλιογραφία για κάτι τέτοιο. Διαπιστώνονται παρόλα αυτά κάποιες δυσκολίες και εμπόδια στην διαμόρφωση συνενέσεων και συμφωνιών. Ενώ και στις δύο υδάτινες λεκάνες στη συνένεση στηρίζεται η συνεργασία. Βέβαια υπάρχουν σημαντικές πρόοδοι σε θέματα περιφερειακής συνεργασίας και ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ε, τα τελευταία επιτεύγματα της ICAT, της οργάνωσης δηλαδή που διαχειρίζεται την αλία του τόνου ενό είδου με ιδιαίτερα έντονες μεταναστευτικέ τάσει. Επίσης έχουμε την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο τη θάλασσα και τις ε, κρατικές, ε, διακρατικές συνεργασίες που είτε έχουν διμερεί, είτε υποπεριφερειακό, είτε περιφερειακό χαρακτήρα. Κατά τη γνώμη μου, οι διμερείς συμφωνίες μπορούν ε, να θεωρηθούν ως συμπληρωματικές για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έχουμε πολλά παραδείγματα όπου η σύναψη διμερών συμφωνιών θα ήταν η καταλληλότερη λύση. Τώρα, ποια είναι τα πλονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τα υπέρ και τα κατά της περιφερειακής συνεργασίας. Υπάρχουν ε, πολύ σημαντικά επιχειρήματα υπέρ της ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας. Γιατί σε μια ολοκληρωμένη ελευτική πολιτική, ευρωπαϊκή ελευτική πολιτική, είναι σημαντικό να δώσουμε έμφαση στην περιφερειακή προσέγγιση, στην περιφερειακή εστίαση. Είχαμε πολύ σημαντικές πρόοδους ε, στην ε, θαλάσσια διακυβέρνηση και στον χωρικό προγραμματισμό. Όλα αυτά εντάσσονται στην περιφερειακή προσέγγιση, στην περιφερειακή έμφαση που δίνουμε. Βέβαια αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν στην πορεία αυτή, σε αυτή την ε, περιφερειακή, δηλαδή και υποπεριφερειακή προσέγγιση. Βέβαια, οι τελευταίες τάσεις και οι τελευταίες πρωτοβουλίες για τη διαχείριση των κοινών πόρων και περιλαμβάνουν τη ελεία ως τη της θαλα... διαχείρισης θάλασσας, όλα αυτά εντάσσονται σε ένα πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας. Τέλος, η έκθεση περιλαμβάνει και μία ντουζίνα περίπου, δώδεκαρια συστάσεων. Θα ήθελα να τις συνοψίσω σε πέντε σημεία που παρουσιάζω στη διαφάνεια αυτή, αλλά υπογραμμίζω ιδιαίτερα την υποπεριφερειακή διάσταση. Θεωρώ ότι η υποπεριφερειακή αυτή διάσταση προσαρμόζεται καλύτερα στις οκενογραφικές πολιτικές και δικαιοδοτικές συνθήκες. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Μεσογείου. Αυτά προς το παρόν, αυτά από μέρους μου και σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά, κύριε Σουάρες Ντεβιβέρο. Θα δώσω τώρα το λόγο στον τελευταίο μας καλεσμένο, τον δόκτωρα Κάντι, για να μας κάνει τη δική του παρουσίαση. take Oh, oh, uh, Ωραία. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε μια ιδιαίτερη πτυχή της Μεσογείου που είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Είναι πάρα πολύ ρηχή η υφαλοκρηπίδα, μάλλον είναι πολύ στενή η υφαλοκρηπίδα στα περισσότερα μέρη της ε, της ε, Μεσογείου, στον κόλπο της Λιών και στην Αδριατική γενικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα αλία σε μικρό βάθος, αλλά στα περισσότερα μέρη είναι μεγάλο το βάθος της ε, Μεσογείου. Και αν δείτε, το όριο των 50 μιλίων από την ακτή μπορεί να μην έχει νομική βάση αυτή, αυτός ο διαχωρισμός, αλλά η περισσότερη αλληλεία λαμβάνει η χώρα σε απόσταση μέχρι 50 ναυτικών μιλίων από την ακτή, γιατί πιο επέκεινα αυτού του ορίου είναι πολύ μεγάλο το βάθο τη θάλασσα. Αυτό είναι ένα λόγο για τον οποίο είναι ενδιαφέρον να δούμε την διαχείριση τη Μεσογείου και όχι απλώ να με διαφορετικό τρόπο και όχι να γενικεύουμε απλώ από τι διατάξει που ισχύουν στη Βόρεια Θάλασσα που είναι τελείω διαφορετική η υδατογραφική κατάσταση. Πρέπει να δούμε λοιπόν αυτή την κατάσταση, τη διαφορετική της Μεσογείου, πρωτού προχωρήσουμε σε πάρα πολλέ προβλέψεις. Όταν λοιπόν μιλήσω για την πτυχή του ασύλου κατά κάποιο τρόπο για, τα, για τους ηχθείς, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από αυτή την άποψη. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι δεν έχουν διακηρύξει ΑΟΣ οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες όλες τις χώρες Μεσογείου, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και μια διαχείριση για την ανοιχτή θάλασσα. Δεν έχω δεν είχα τον καιρό να ελέγξω απόλυτα όλα αυτά τα στοιχεία που σας αναφέρω και εγώ είχα συντάξει αυτή την έκθεση το Σεπτέμβριο και έκανα ορισμένε βελτιώσεις μετά από τα στοιχεία που πήρα σε σχέση με τη Μεσόγειο. Αν θέλετε λοιπόν να ελέγξετε μερικά από αυτά τα στοιχεία περαιτέρω, αυτό θα είναι χρήσιμο. Υπήρξε πρόβλημα, όπω ξέρετε, στο να καταλήξουμε σε ένα κοινό αλλιευτικό πλαίσιο, όπω ανέφερε και ο προηγούμενος ομιλητής. Σε πολλέ περιπτώσεις υπήρξε έλλειψη οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων που επηρέασε αυτό από πολλές χώρες. Επομένως υπήρχε μια μείωση τη συμμετοχή του σε αυτήν την αλλιευτική πολιτική και τη διαχείρισή τη, Έχουν προταθεί στο Συμβούλιο Αλίας στη Γενική Επιτροπή Αλία για τη Μεσόγειο συγκεκριμένα, υπήρξαν πολλές ιδέες οι οποίε έχουν διατυπωθεί. Η μορφή που έχει τώρα η Επιτροπή για την Αλία στη Μεσόγειο φαίνεται σε αυτό το γράφημα. Στο κέντρο είναι η Κομισιόν, στην οποία υπόκειται η Επιστημονική Επιτροπή και ορισμένες υποεπιτροπές που αφορούν την ε, εκτίμηση των ε, αλλιευμάτων, στατιστικές και πληροφορίες, οικονομικές και κοινωνικές ε, επιστήμες, θαλάσσιο περιβάλλον και επίσης το θέμα της ιχθυοκαλλιέργειας. Ε, Είναι η μόνη τέτοια επιστημονική επιτροπή στον κόσμο, ίσως που ασχολείται με την ηχθειοκαλλιέργεια και αυτό τροποποιεί σημαντικά την προσέγγιση, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά που γίνουν μέσα στα 12 και μόνο ναυτικά μίλια από την ακτή. παρά το γεγονό ότι αυτό είναι μια καθαρά εθνική ζώνη, οι περισσότερε δραστηριότητε ηχθειοκαλλιέργεια περιορίζονται εκεί. Από την άλλη πλευρά έχουμε την συνεργασία με την ε, ICAT, που, υπάρχει, που είναι η αρμόδια επιτροπή για τον τόνο και διάφορες ομάδες εργασίας για τα είδη μεγάλου βάθους, τα πελαγικά κτλ. αριστερά έχουμε τις υποπεριφερειακές ε, οντότητες του ΦΑΟ που συνεργάζονται με την Επιτροπή για την Αλία στη Μεσόγειο. Ένα από τα προβλήματα τώρα που γίνεται σαφές και αυτό φάνηκε από την έκθεση του κύριου Μακόαερ που έκανε μια α, πρώτη, μια πρώιμη έκθεση για τα θέματα αυτά είναι ότι όταν φεύγουμε από τις περιοχές οι οποίες βρίσκονται στην βορειοδυτική Μεσόγειο και προχωρούμε προς τα ανατολικά, οι πόροι μειώνονται σε σχέση με πληροφορίες και έχουμε πάρα, πολλά, πάρα πολύ λίγα στοιχεία από τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα λοιπόν, ένα πρόβλημα όμως το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα. Τώρα, αν βελτιώνται τα επιστημονικά στοιχεία που συλλέγουμε ή όχι. Το γεγονός ότι έχουμε ένα αριθμό επιμέρους φορέων που ασχολούνται για τα θέματα αυτά, αυτό δεν έχει οδηγήσει σε υψηλό όγκο δεδομένων και καλύτερη τεχνική ανάλυση. Σε πολλές περιπτώσεις οι τεχνικές διαδικασίες είναι ακόμα υπό διευκρίνηση στις αντίστοιχες επιτροπές. Έχουμε μια πολύ καλή ιστοσελίδα βέβαια και υπάρχουν πολλές πληροφορίες που μπορεί κανείς να αποκομίσει από εκεί και πολλές συστάσεις για τη διαχείριση έχουν προκύψει από μέρημνα για την προστασία των αλληλευτικών ειδών και αναφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα. Τώρα, λίγε, λίγα από τα 51 ουσιαστικά, ουσιαστικής σημασίας θαλάσσια είδη καλύπτονται από συστάσεις. Το να το κάνουμε αυτό κάθε χρόνο για όλα τα σημαντικά είδη, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι ε, βιώσιμες οι συστάσεις ανά είδος για τον έλεγχο της αλληλευτικής ε, προσπάθειας και για τις ποσοστώσεις. Και το θέμα του περιορισμού της προσπάθειας είναι το πιο σημαντικό για τη Μεσόγειο. Αλλά το να έχουμε τρεις ή τέσσερις αξιολογήσεις για τα αλλιευτικά είδη το χρόνο θα ήταν, αναπεριοχή θα ήταν πολύ σημαντικό στόχος να επιτύχουμε. Καταρχήν όμως θα πρέπει να έχουμε ένα πιο απλό τρόπο αντιμετώπισης με μελέτες που δείχνουν το αποτέλεσμα της αλίευσης και την ε, για την αλία με που φυσικά αλλιεύουν πολλά είδη, επομένως να γίνονται μελέτες επί τη βάση των αλλιευμάτων από τράτες που καλύπτουν ιδιαίτερα, που καλύπτουν πολλά είδη ηχθείων. Και αυτό συμπληρώνει τις μελέτες για συγκεκριμένα είδη που αναφέρονται από τις μελέτες. Κάποιες μελέτες λοιπόν έχουν γίνει από την Επιτροπή, άλλες έχουν γίνει από τη STEF, αλλά όλα αυτά δεν επαρκούν για μια πλήρη διαχειριστική προσέγγιση. Έχετε τώρα ένα διάγραμμα, ένα γράφημα που παρουσίασε το 2010 ο Φερούγιο. Από τότε τα πράγματα έχουν αλλάξει σημαντικά. Κάτι το οποίο με εντυπωσιάζει είναι το πόσο γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα. Το τελευταίο καιρό κάποια από αυτά που θα πω ίσως είναι πεπαλαιωμένα ίσως ως πληροφορίες. Γι' αυτό έχω κάνει κάποιες αλλαγές στο έγγραφό μου που εμφανίζεται μόνο στο διαδίκτυο. Βλέπετε εδώ ότι έχουμε πολύ λίγα, πολύ λίγα στοιχεία για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα υπάρχουν κάποια στοιχεία από την Αίγυπτο και την Κύπρο και στην Μαύρη Θάλασσα. Δεν είναι σωστό ότι δεν υπάρχουν καθόλου αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις, οι πρώτες είχαν γίνει το 1970 από τις ε, επιτροπές τότε επικομμουνιστικού καθεστώτος στις χώρες αυτές επί τη βάση μιας τεχνολογίας που ήταν στα ίδια επίπεδα με τη τεχνολογία που χρησιμοποιούταν στο Βόρειο Ατλαντικό. Η συλλογή λοιπόν και η αξιολόγηση στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα είναι το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την διαχείριση. Υπάρχουν στοιχεία τα τελευταία πέντε ή τέσσερα χρόνια η προσπάθεια, η αλληλευτική που ασκείται έχει μειωθεί σημαντικά. Αυτό πράγματι έχει λάβει χώρα, αλλά δεν υπήρξε μια αντίστοιχη αύξηση στην αυθονία των αλληλευτικών ειδών. Η Επιτροπή λοιπόν για την ε, Αλία στη Μεσόγειο θα πρέπει να αποφύγει μια κατάσταση όπως αυτή που ισχύει σήμερα, όπου κάθε περιοχή αντιμετωπίζεται μεμονωμένα από μια χωριστή υποεπιτροπή. Πρέπει να ενσωματώσουμε καλύτερα τις δραστηριότητες αυτών των υποεπιτροπών. Θα πρέπει να συναντιόνται συγχρόνως σε αιτήσιο επίπεδο και να συνεργάζονται ή όχι. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το συζητήσουμε. Επίσης, η μέθοδη ανάλυσης δεδομένων για στόχους διαχείρισης. οι απλές μέθοδοι που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση θα μπορούν να είναι επαρκείς για μια διαχείριση επί τη βάση της αρχής της πρόληψης. Μια υποεπιτροπή επίσης για την παρακολούθηση της ε, περιβαλλοντικής αλλαγής που είναι πολύ σημαντική για τη Μεσόγειο θα πρέπει και αυτή να προτείνει τον αποκλεισμό συγκεκριμένων ε, περιοχών σε παρασυρώμενα αλλιευτικά είδη και να ρυθμίσει την απόρριψη αλλιευμάτων. Ο κύριος Σπανιόλο περίγραψε, περίγραψε ορισμένα θέματα που άπτονται της, ε, των κοινωνικών και οικονομικών πτυχών. Είναι γνωστό ότι λόγω της χαμηλής παραγωγικότητας Μεσογείου κυριαρχούν τα μικρά ψάρια στην αγορά, μικρή παραγωγικότητα και μεγάλη υπερεκμετάλλευση. Αλλά υπάρχει και μία παράδοση του να ε, έρχονται τα, πιά, ψάρια υπομορφή μικρών νυχτίων στο πιάτο. Και αυτό ιδίως στις κύριες τουριστικές περιοχές της Μεσογείου. Πολλοί τουρίστες πηγαίνουν εκεί και περιμένουν να δοκιμάσουν παραδοσιακά ε, ψαροφάγια, ε, γεύματα που περιέχουν ψάρια και πολλές φορές αυτά απαρτίζονται και από μικρά ψαράκια. Και είναι αδύνατο να πάψει να γίνει τα αυτών των ειδών. Η, το κλείσιμο ορισμένων περιοχών αλίας είναι μια μορφή διαχείρισης για την ε, διαχείριση από τη βάση πολλαπλών ειδών και η διαδικασία των TERFs επίσης έχει αναφερθεί. Εγώ θέλω να σας αναφέρω εδώ πέρα τα διαγράμματα ε, κύκλου ζωής για τρία είδη ηχθείων που έχουν παρουσιαστεί καταρχήν στη 1960 έχουν κάπως λησμονηθεί αυτά τα στοιχεία αλλά φαίνεται ότι βρίσκονται στην ε, άκρη της υφαλοκρηπίδας στα θαλάσσια αυτά είδη πηγαίνουν σε περιοχές ε, αναπαραγωγής κοντά στην υφαλοκρηπίδα ή πάνω στην υφαλοκρηπίδα και τελικά κυκλοφορούν προς τα βαθύτερα ύδατα. Στα αβαθή ύδατα η αλία με την τράτα σε μεγάλο βαθμό ε, εκμεταλλεύεται και τους γόνους ή τα ψάρια τα οποία είναι σε φάση ε, αναπαραγωγής. Αυτό είναι το λεγόμενο υπόδειγμα refugium και στην δεκαετία του 1980-1990 παρά το γεγονός ότι υπήρχε μεγάλη, ε, μεγάλος έλεγχος για τις στράτες συνέχιζε να υπάρχει αλία νεαρών ηχθείων, χωρίς κανένα έλεγχο. Πολλά λοιπόν από τα, όπως σας είπα, είναι βραχώδης η περισσότερη φαλοκρηπίδα της ε, Μεσογείου και επομένως όχι εύκολα ε, εκμεταλλεύσιμη. Το γεγονός ότι γίνεται αυτή η χρήση τρατών ε, πάνω από βαθύτερα ύδατα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει την διατήρηση της έννοιας του ρεφούγιου, δηλαδή του να μπορούν να υπάρχουν χώροι όπου η αναπαραγωγή των ηχθείων γίνεται απρόσκοπτα. Και η εφαρμογή αυτής της αρχής έχει αρχίσει να, ότι πρέπει να υπάρχει το refugium αρχίζει να εφαρμόζεται στον κόλπο της ε, στον ε, κόλπο της ε, Τουλώνος. Και για, για ορισμένα είδη γάδου ιδίω ισχύει αυτή η μορφή περιορισμού. Νομίζω ότι αυτή θα είναι και η καλύτερη λύση για να επιλυθούν όλα αυτά τα προβλήματα για την προστασία των ε, νεαρών ηχθείων. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια, ένα κλείσιμο ορισμένων περιοχών σε αλλιευτικά είδη τα οποία ε, φτάνουν μέχρι το βυθό και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να υπάρξει προστασία των χώρων, των περιοχών αναπαραγωγής και ε, της ανάπτυξης των νεαρών ηχθείων. Εδώ και ένα, εδώ και ένα αιώνα περίπου οι τράτες ε, ε, στην ακτή της Ισπανίας έχουν αρχίσει να αναζητούν γαρίδες σε περιοχές μέχρι 800 μέτρα βάθους. Και είναι σαν οργωμένο χωράφι πια ο βυθός της θάλασσας στις περιοχές αυτές. Αυτό οδηγεί στο να υπάρξουν ζήματα τα οποία μεταφέρονται σε βαθύτερα ε, σε μεγαλύτερα βάθη και αυτό αλλάζει και την κατανομή των θαλασσίων ειδών. Και εδώ έχετε ένα παράδειγμα από τις ΗΠΑ όπου έχει απαγορευτεί η χρήση των αλυσίδων στις στράτες και βλέπετε μια α, μαύρη περιοχή που είναι η βραχώδης αυτή η περιοχή και βλέπετε τι προέκυψε όταν υπήρξε η απαγόρευση της χρήσης αλυσίδων στις ε, τράτες, ώστε με την εφαρμογή αυτού του κανόνα μειώθηκε σημαντικά η καταστροφή που παράγεται στις ε, βραχώδεις περιοχές και η καλύτερη προστασία των νέων νυχθείων. Η προστασία των νέων νυχθείων μπορεί να γίνει επίσης με το να μειωθεί η εποχική προσπάθεια σε περιοχές όπου γίνεται η εκόλαψη και η ανάπτυξη των νεαρών νυχθείων. Οι μελέτες για την επιβίωση των νεαρών νυχθείων σε... που, που περνάνε μέσα από τα μάτια των δικτύων για γάδο στο Βόρειο Ατλαντικό, έδειξαν ότι υπάρχει και φυσιολογικό στρες στους ηχθείς που επιβιώνουν. Στη συνέχεια όμως έχουν μεγαλύτερους ρυθμούς θνησιμότητος από τους ε, θηρευτές τους. Επομένως, η σημασία της αύξησης του μεγέθους των ματιών δεν είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζαμε. Εδώ έχουμε ένα ε, γράφημα που δείχνει ένα, μια αντιμετώπιση διαχείρισης που έχει ευρύτερο χωρικό χαρακτήρα. Εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την σχέση μεταξύ χθιοκαλλιέργειας, τουρισμού και αλίας. Εδώ σας δείχνω ένα υποθετικό διά, διάγραμμα όπου υπάρχει μια ζώνη ρεφούγιου, υπάρχει μια ζώνη όπου μπορεί να γίνεται χρήση τρατών και υπάρχουν επίσης περιοχές όπου δεν επιτρέπεται να υπάρχουν τράτες κοντά στην ακτή. Είναι περιοχές όπου εκολάπτονται οι νεαροί ηχθείες και περιοχές όπου υπάρχουν χώροι μονάχα για καλλιέργεια. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας λοιπόν ένα τέτοιο σχήμα όταν σχεδιάζουμε τα turfs στην περιοχή της Μεσογείου. Και τώρα ερχόμαστε στη σχέση της Επιτροπής με τη Μεσόγειο και του Εύξηνου Πόντου. Δεν θέλω να πω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά στην δεκαετία του 1990 υπήρξε μια κρίση η οποία προέκυψε από τις εκροές ε, θρεπτικών ουσιών από τον Δνήπερο και τον Δούναβι και από την Μέδουσα μνε, Μνεμιόψης που μπήκε στη Μαύρη Θάλασσα από έκπληση δεξαμενών πλοίων που προχώρησαν από τις Αμερικανικές ακτές. Το αποτέλεσμα ήταν ότι υπήρξε μεγάλη κατανάλωση ζωοπλακτών, ε, αυγοτάραχου και νέων, ε, νέων ηχθείων, ώστε να μειωθεί σημαντικά η αλίευση πελαγικών ηχθείων στη δεκαετία του 90 και σε ε, μείωση οξυγόνου στην περιοχή αυτή εφόσον καταναλώθηκε από αυτά τα αυτά τις θερευτικές μέδουσες ένα μεγάλο μέρος του οξυγόνου. Όλο αυτό έχει αλλάξει σημαντικά τη μορφή της Μαύρης Θάλασσας και έχει κάνει τις προηγούμενες μελέτες σε σχέση με την Μαύρη Θάλασσα ουσιαστικά άσχετες με την τωρινή διαχείριση των ηχθείων της Μαύρης Θάλασσας. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν μερικές σημαντικές χώρες στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου που δεν είναι μέλη της Επιτροπής για τη Μεσόγειο. Και εδώ έχουμε δύο δυνατές ε, επιλογές, είτε να έχουμε ένα αυτόνομο σώμα διαχείρισης για τον Ευξήνο Πόντο ή δεύτερον να πείσουμε τις χώρες αυτές να γίνουν μέλη της Επιτροπής για τη Μεσόγειο. Εγώ πιστεύω θα πρέπει να υπάρξει και ένα χωριστό πάνελ της Επιτροπής για τη Μεσόγειο για τα θέματα αυτά, γιατί το να συνδυάσουμε την Επιτροπή για τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο λόγω τη διαφορετική μορφή των δύο θάλασσών και χαοτικού χαρακτήρα. Θα έπρεπε λοιπόν να σκεφτούμε να έχουμε δύο χωριστά πάνελ. Επομένω, πιστεύω ότι η GFCM, η Επιτροπή για τη Μεσόγειο, έχει πολλέ επιτροπέ. πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται σε πολυδιάστατα θέματα. Θα πρέπει να βρουν μια λύση για το να μπορούν να συμμετέχουν και οι μικρότερε χώρε. οι, οι που έχουν περιορισμένη οικονομική σημασία της αλίας και κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε και τη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για διαχειριστικές συναντήσεις ή άλλες μορφές συναντήσεων. Πώς η SDCF e θα μπορέσει να συμπληρώσει το έργο της Επιτροπής για την Μεσόγειο και των αξιολογήσεών τους θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. Και επίσης η στατιστική προσέγγιση είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί. Χρειαζόμαστε περαιτέρω να έχουμε σημεία αναφοράς οριακού χαρακτήρα. Η Επιτροπή για τη Μεσόγειο μου είπε ότι έχουν προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Τα σημεία αναφοράς οριακού χαρακτήρα σημαίνουν ότι το επίπεδο αυθονίας των νυχτίων πέφτει κάτω από ένα αποδεκτό ε, επίπεδο ή εάν υπάρξει μια ε, ε, μείωση κάτω από το ελάχιστο επίπεδο. Επίση, είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε τι χώρε σε τοπικό επίπεδο για την εφαρμογή των συστάσεων τη Επιτροπής για τη Μεσόγειο. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για να συμπληρωθούν οι προσπάθειε. Η συνεργασία με εξωτερικού φορεί για την εφαρμογή περιβαλλοντικών ρυθμίσεων επίσης φαίνεται ότι είναι κατάλληλη στα πλαίσια αυτά. Το να κλείνονται ορισμένες περιοχές, να αποκλείονται από την αλληλεία είτε εποχικά είτε μόνιμα, αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη λήψη αποφάσεων και ιδίως η Επιτροπή για την Ιχθειοκαλλιέργεια θα πρέπει να συνεργάζεται με τοπικές αρχές που έχουν τέρφ, έχουν τοπικά δικαιώματα χρήσης η αύξηση στο, μάτι στο μέγεθος του ματιού των δικτών θα πρέπει να αντιμετωπίσετε προσεκτικά γιατί υπάρχει άμεση πρόκληση θρησιμότητα από τις στράτες ακόμα και για αυτά τα ψάρια τα οποία επιβιώνουν μέσα από τα δίκτυα. Και επομένως όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε συνολικά. Και επίσης θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στη σημασία της, ε, να δώσουμε σημασία στην οικονομικές πτυχές, όχι με στόχο να έχουμε απλώς το μεγαλύτερο τονάζ αλλιευμάτων, αλλά να έχουμε την, την μεγαλύτερη αξία των αλλιευμάτων. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε καλύτερα ποια είναι η τοπική ζήτηση στη Μεσόγειο για διάφορες μορφές ηχθείων. και να προσαρμόσουμε τις μορφές αλίες σε αυτό το σχήμα ζήτησης. Επίσης η προσέγγιση Refugium που υπογραμμίστηκε εδώ, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κλείνουμε ορισμένες περιοχές στις υφαλοκρηπίδες που έχουν βραχώδη πυθμένα στην ε, αλία για να προστατεύσουμε τους νεαρούς ηχθείς. Το να μειώσουμε λοιπόν την χρήση τρατών σε περιοχές Refugium, αυτό είναι μια λύση αλλά επίσης μπορούμε να έχουμε και απαγόρευση σε τροποποίηση των κρατών που τους επιτρέπουν να λειτουργούν σε βραχώδεις πυθμένες. Χρειαζόμαστε όταν υπάρχει περίφραξη κάποιου, κάποιου χώρου να υπάρχει και παρακολούθηση από δορυφόρους από τους, ε, της στράτας και με άλλες μεθόδους και να υπάρχουν οι κατάλληλε κυρώσει. Και τέλο, χρειαζόμαστε να έχουμε μια διάγνωση τη κατάσταση των αλληλευτικών αποθεμάτων αλλά και των ηχθειοτόπων και γενικά η χρήση των τρατών δεν βοηθάει την προστασία των ηχθειοτόπων. Η εφαρμογή των, των συστάσεων τη ΣΑΚ και τη Επιτροπή είναι πάρα πολύ σημαντική για τη σωστή διαχείριση και όλα αυτά εξαρτώνται φυσικά και από τη δράση των κρατών μελών για να εφαρμόσουν τι συστάσει τη GFCM, τη Επιτροπή για τη Μεσόγειο. Θα ήθελα εν κατακλείδη να σας πω ότι ίσως οι κρίσεις που αναφέρονται εδώ πέρα είναι υπερβολικά αυστηρές σε σχέση με αυτό το οποίο έχει γίνει στη Μεσόγειο και η Επιτροπή για τη Μεσόγειο πιστεύω έχει κάνει κάποια αρκετά επιθετική δουλειά τα τελευταία δύο χρόνια και θα πρέπει να προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής στην για τη Μεσόγειο για την εφαρμογή όλων αυτών των συστάσεων της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κάντι. Ακούσαμε λοιπόν τους τρεις εμπειρογνώμονές μας. Θα ακολουθήσει γύρος ερωταπαντήσεων. Ποιος θέλει το λόγο, κυρία Λέβιν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους ε, καλεσμένους μας. Εγώ κατάγομαι από χώρα του Βορρά και πραγματικά ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ενημέρωση για την Αλία στη Μεσόγειο. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, της ρύθμισης της αλίας στη Μεσόγειο σε σχέση με την αλία στη Βόρεια τη Βαλτική θάλασσα. Κάτι που με εντυπωσίασε, γι' αυτό και θα ήθελα να θέσω και μια σχετική ερώτηση, είναι το θέμα της ανοιχτής θάλασσας στη Μεσόγειο. Γιατί αναφέρθηκε ότι το ποσοστό της ανοιχτής θάλασσας, πέραν των χωρικών υδάτων δηλαδή, έχει μειωθεί τον τελευταίο καιρό. Από το 40% στο 30%. Πώς θα μπορούσατε να μας το αναλύσετε Δηλαδή υπάρχουν χώρες που διεκδικούν ε, ΑΟΣ, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Τι γίνεται, γιατί έχει μειωθεί αυτό το ποσοστό της ανοιχτή θάλασσας στη Μεσόγειο. Πολλές φορές ασχοληθήκαμε με τον εύξηνο πόντο και έχω την αίσθηση ότι καλύτερο θα ήταν να έχει ξεχωριστεί η Επιτροπή η, Μεσο... η Μαύρη Θάλασσα από το να υπαχθεί στην Γενική Επιτροπή της Αλίας για τη Μεσόγειο. Ποια είναι η δική σας γνώμη πιστεύετε ότι χρειάζεται ε, ειδική επιτροπή η Μαύρη Θάλασσα ή όχι. Και κάτι που με κατέπληξε κάπως, γιατί ήταν κάτι πρωτότυπο, δεν το έχω ακούσει, είναι ότι αυξάνεται το, θα αυξηθεί η θνησιμότητα των ψαριών αν αυξηθεί ε, το εύρος των ματιών των ε, τρατών. Δεν κατάλαβα καλά, επειδή περνώντα από τα μάτια, παρόλα αυτά, λόγω του στρες, θα αυξάνεται η θνησιμότητά τους, οπότε δεν εξυπηρετεί η διεύρυνση των ματιών. Και επίσης, τι γίνεται με τις προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές, δηλαδή τις περιοχές εκτός των αλληλευτικών πεδίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λέβιν. Άλλος κανείς? Ωραία, ας ακούσουμε τους καλεσμένους μας τώρα. Ο κύριος Κάντι πρώτα. Εκτός μικροφώνου ο κύριος Κάντι. Το τελευταίο ερώτημα της έμεσης νησιμότητας. Έγινε πολλή δουλειά στη Σκωτία και στις σκανδιναβικές χώρες για το θέμα αυτό. Και αυτό που με εξέπληξε είναι ότι αυτή η δουλειά δεν έχει ληφθεί υπόψη από αυτούς που εξεργάζονται τα αποθέματα. Έγιναν πειράματα. Συλλέγεται ο γόνος αφού συλληφθεί από το δίχτυ, μένει σε κλωβούς και μελέτησαν πόσοι επέζησαν. Και μεγάλο ποσοστό του γόνου δεν επέζησε. Γιατί. Έχουν περιορισμένου ε, περιορισμένους ενεργειακούς πόρους στο σηκώτη τους. Εάν επί μισή ώρα ε, κορυμπούσαν μπροστά από το δίχτυ και μετά περάσουν από το δίχτυ δεν σημαίνει ότι επέζησαν. Και υπάρχει και άλλη πτυχή. Σε πολλές περιπτώσεις οι εμπορικές στράτες ε, ψαρεύουν και σέρνουν τα δίχτυα πάνω από την ίδια περιοχή πολλές φορές. Οπότε τα ψάρια μπορούν να έχουν περάσουν σε μια μέρα να έχουν περάσει πολλές φορές από το δίχτυ. Δεν τα αναζωογονεί όπως καταλαβαίνετε τα ψαράκια. Μπορεί να εκπαιδεύονται στο κολύμπι, να γίνονται καλοί κολυμβητές, αλλά δεν είναι καλό για τα μικρά ψαράκια και πολλοί γόνοι βρίσκονται σε περιοχές με ε, χλωρίδα ε, και αφαιρείται η χλωρίδα από την περιοχή που ζουν και δεν μπορούν να φάνε. Άρα, άμα έχει βλάστηση ο βυθός, δεν ψαρεύουμε εκεί. Δεν έχουν τα φάντα τα ψάρια μετά. Και πρέπει και να γλιτώσουν τα ψάρια που φτάνουν στη, στο μέγεθος αναπαραγωγής. Ε, και βλέπει κανείς καμιά φορά ότι στα δίχτυα δεν υπάρχουν ε, ε, μη γόνοι και πρέπει να τη γλιτώσουν για να μπορέσουν να γεννήσουν. Αν αλλιεύεις στο βάθος και ε, ψαρεύεις μπακαλιάρο ή γαρίδα, δεν βοηθάς την παράκτεια. Είτε έχεις μάτι 40 χιλιοστά ή άλλο μέγεθος, δεν είναι το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα είναι τι κάνεις στο οικοσύστημα από το οποίο εξαρτάται το ψάρι. Το πραγματικό σφάλμα στους υπολογισμούς, όπου βλέπουν βελτιωμένη απόδοση με την αύξηση του ματιού του δικτυού, είναι ότι στους υπολογισμούς δεν λαμβάνουν υπόψη το 20% και παραπάνω που σκοτώνεται κατά τη διάρκεια ε, του ψαρέματος ε, με αυτόν τον τρόπο. Ε, μπορεί να είναι μεγαλύτερο το μάτι, ε, δεν βελτιώνει όμως την απόδοση. Μπορούμε να πιάσουμε μικρή γαρίδα, μικρά κεφαλόποδα και είναι άκρος πολύτιμα αυτά τα είδη. Ένα-δύο εκατοστά μήκος έχουν. Και όπου πας εστιατόριο στη Μεσόγειο μπορείς να φας ένα πιάτο με μικρές γαρίδες, μικρά καλαμάρια, μικρά ψάρια και είναι παραδοσιακός τρόπος κατανάλωσης ψαριού σε αυτές τις χώρες. Αν αυτά τα ψάρια, τα νέα ψάρια, κοστίζουν στην αγορά περισσότερα ένα κιλό από τα μεγάλα και αν πας ιταλικά εστιατόρια ούτως ή άλλως δεν θα βρεις συχνά α, ε, ε, φιλέτα ψαριού, βρίσκεις ψαράκια στο πιάτο είναι θέμα συνήθεια, Αυτό τρώνε οι άνθρωποι. Άρα πρέπει να, να δει κανεί και την κοινωνικο-οικονομική ζήτηση για κάποιο είδο. Όχι τη βιομάζα απλώς του υπολογισμού. Χρησιμοποιείται πολύ απλουστευμένη μέθοδος για την αξιολόγηση των αποθεμάτων. Πρέπει να σκεφτούν και άλλες ε, Βιολογικέ περιβάλλοντο, περιβάλλοντος, οικονομικέ. Μάλιστα. Άλλος κανείς? Eh, Ο κύριος Σουάρες Δεβιβέρο. Θα ήθελα να διευκρινίσω μόνο την ορολογία που χρησιμοποιούμε. Όταν μιλούμε για αλληλεία ανοιχτή θάλασσα. Στην περίπτωση της Μεσογείου, Πολλές φορές η ανοιχτή θάλασσα <laughs> είναι κοντά. Δεν σημαίνει ότι κανείς ε, ξανοίγεται πολύ μακριά για να ε, αλλιεύσει σε ανοιχτή θάλασσα. Αν δούμε το χάρτη με τις δικαιοδοσίες, και ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα, οποιοδήποτε σκάφος που ξεπερνάει, απομακρύνεται 12 μίλια από την ε, ακτή, βρίσκεται ήδη στην ανοιχτή θάλασσα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αλλιεύει, ότι πραγματοποιεί αλληλεία ανοιχτής θάλασσας. Οπότε θα πρέπει ίσως να αναθεωρήσουμε την ορολογία που χρησιμοποιούμε και να χρησιμοποιήσουμε άλλους δείκτες στην περίπτωση αυτή. Εγώ προσπάθησα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον, θα μειωθεί το ποσοστό, δραστικά το ποσοστό της ανοιχτή θάλασσας του τμήματος δηλαδή που δεν εμπίπτει στα χωρικά ύδατα. Οπότε και ο τρόπος δια, διαχείρισης θα πρέπει να τροποποιηθεί. Ε, έτσι θα επηρεαστεί και ο ρόλος ε, κάποιων ε, επιτροπών ή οργάνων, όπως η Γενική Επιτροπή επιτροπη αλλιες για τη Μεσόγειο. Γιατί όπως είδαμε και σε άλλες εκθέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακόμη και δεν υπάρχει ε, ανοιχτή θάλασσα, ακόμη και μειώνεται το ποσοστό, θα είναι σημαντικός ο ρόλος αυτών των ε, οργάνων. Βέβαια, παρόλο που υπάρχει ανοιχτή θάλασσα, έστω και 30%, το υπέδαφος του πυθμένα της Μεσογείου ε, υπόκειται στην εθνική τη δικαιοδοσία. Δηλαδή όλα τα είδη τα βενθικά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα μίας από τις παράκτιες χώρες. Ώστε για να ασκηθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα στο, στην υφαλοκρηπίδα δεν χρειάζεται να διεκδικηθεί με νόμο σε αντίθεση με αυτό που ισχύει για τις ε, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες με τις αλληλευτικές ζώνες ή τις ζώνες ε, οικολογικής προστασίας. Ευχαριστώ. Έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Γκαρθία Γέρρο. Ευχαριστώ. Δύο λόγια μόνο, γιατί ήθελα να κάνω ακριβώς αυτή την ερώτηση στον καθηγητή Σουάρης Δεβιβέρο, γιατί πολύ συχνά ακούμε από τους ευρωβουλευτές ε, ακούμε μάλλον πολλές έννοιες που μερικές φορές τις ηχαίωμα στο μυαλό μας. Ε, αλία ανοιχτή θάλασσα δεν ισοδυναμεί κατά με την βιομηχανική αλία. Θα πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Η βιοτεχνική αλία μικρής κλίμακας ε, ή η αλία οστρακοειδών όταν είναι πολύ χρονικά περιορισμένη, μπορεί να τυχει, θα πρέπει να τύχει ειδική θέση στην ε, μεταρρύθμιση τη κοινή ελεύθερη πολιτική και ίσω να προβλεφθούν και ξεχωριστά κονδύλια για την αλία μικρή κλίμακα την παράκτη αλία που είναι πολύ σημαντική ιδιαίτερα για τη Μεσόγειο. Για να μην ε, συνεχιστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει ήδη από οικονομική, ε, οικονομική άποψη και από άποψη απασχόλησης. Γι' αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας. Δηλαδή, έχετε στοιχεία, γιατί είπατε ότι ήδη υπάρχουν πολλές επιστημονικές ε, μελέτες, έρευνες, αξιολογήσεις από τα κράτη-μέλη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε στοιχεία για το επίπεδο ε, της αλληλευτικής ε, ε, ικανότητας, γιατί αναφέρθηκε η λεωνάζουσα αλληλευτική ικανότητα, 80% ανά αλληλευτικό είδος, ε, ανά, αλληλείας, έχετε τελικά στοιχεία. Και σε αυτό το σχέση, στο πλέγμα σχέσεων μεταξύ κρατών μελών μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις τρίτες χώρες, πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε αυτά τα σχέδια αλληλευτικής διαχείρισης. Για να μην έχουμε αυτή την αίσθηση της εγκατάλειψης, γιατί πιστεύω ότι πολύ, πολύ δικαιολογημένα αυτή την αίσθηση έχουν οι αλληλείς από τις τοπικές κοινότητες, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ κύριε Γέρο. Δώσω το λόγο στον κύριο Ντέβις να υποβάλει και τη δική του ερώτηση και μετά μπορείτε να απαντήσετε και στους δύο μαζί. Μια ερώτηση όσον αφορά τα λευτικά αποθέματα. Επί σειρά ετών άκουσα διαφορετικέ αξιολογήσει από καταστροφική κατάσταση μέχρι δεν γνωρίζουμε γιατί δεν έχουμε επιστημονικά δεδομένα. μα λένε ότι υπάρχουν τέτοια επιστημονικά δεδομένα για τη Μεσόγειο και δεν έχουν παρουσιαστεί όλα τα στοιχεία. Την αξιολόγησή σα, Ποια είναι η κατάσταση. Τι ανάγκη υπάρχει για αλλαγή. Αν υπάρχει. Πρώτα ο κύριος Κάντι. Well, ε, Θα έλεγα ότι τα τελευταία έξι χρόνια είδα δραματική αύξηση της γνώσης μας για τα τεκτενόμενα στη Μεσόγειο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ατυχώς, πολύ συχνά η μεθοδολογία που απαιτείται για σωστή αξιολόγηση δεν είναι ανεπτυγμένη πάντα. Υπάρχει, παραδείγματος χάρη, διεθνές, διεθνής μετακίνηση προς αξιολόγηση πολλαπλών ειδών. Αυτές οι μεθοδολογίες όμως δεν έχουν καθοριστεί πλήρω. Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στην κατάσταση όπου ψάχνουμε να βρούμε τα αναγκαία εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε την περιπλοκότητα ενός οικοσυστήματος όπως είναι η Μεσόγειος, που ουσιαστικά μοιάζει ε, με την περιοχή ε, των τροπικών, ε, με τις περιοχές, με Ξέρουμε πολλά περισσότερα από πριν αλλά προσπαθούμε να εισαγάγουμε στη Μεσόγειο μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στο Βόρειο Ατλαντικό και σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι οι ενδεδειγμένες μεθοδολογίες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Αν ξεκινήσουμε με βιοοικονομικό στόχο της αλίας θα καταλήξουμε συντομότερα στην ενδεδειγμένη μεθοδολογία. Ευχαριστώ. Κύριε ή ο κύριος Σπανιόλο, ποιος προτιμάει από τους δυο σας. Σε σχέση με το ερώτημα της κυρίας Κοινοβουλευτικού, έχει δίκιο με την έννοια ότι η βιοτεχνική αλληλεία είναι αυτή η οποία έχει τη μεγαλύτερη σημασία στη Μεσόγειο. Και εν γέννη, η αλληλευτική στόλοι στη Μεσόγειο περιορίζουν την αλία τους μέσα στα εθνικά χωρικά ύδατα. Εκτός από την περίπτωση, και αυτό αφορά κυρίως την ε, Ανατολική Μεσόγειο, που ψαρεύουν πέρα των 6 μιλίων, όπως γίνεται στην περίπτωση της Ελλάδος και της Τουρκίας, επειδή είναι 6 μίλια μάλλον τα χωρικά ύδατα, μπορεί να βρεθούν στην ανοιχτή θάλασσα χωρίς να απομακρυνθούν πάρα πολύ από τους λιμένες τους. τόνισα ότι για τα ιδιαίτερα μεταναστευτικά αλλιευτικά ε, είδη είναι απαραίτητο να αλλάξει αυτό το σχήμα. Γιατί σε αυτήν την περίπτωση έχουμε χώρες οι οποίες δεν είναι παράκτιες, οι οποίες αλλιεύουν αυτά τα είδη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξακολουθεί το μεγαλύτερο μέρος της αλίας στη Μεσόγειο να βασίζεται στη μικρή βιοτεχνική αλία που αλλιεύουν τοπικά σε παράκτιο επίπεδο και με βιοτεχνικά μέσα. Για να κλείσουμε τη συζήτηση, ο κύριος Σπανιόλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκπλήσωμαι κάπως από το ερώτημα του κυρίου Ντέιβις. Ήθελα να το πω και πριν μάλιστα αυτό. Υπάρχει Υπάρχουν στοιχεία. Το πρόβλημα είναι να χρησιμοποιηθούν οι διαθέσιμες πληροφορίες. Και να ξέρει κανείς αν υπάρχουν που υπάρχουν. Τα τελευταία χρόνια, δεν θέλω να αναφερθώ στα περασμένα 500 χρόνια, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει τέτοια αλληλεξάρτηση μεταξύ των επιστημόνων στην Ευρώπη, όχι μόνο ε, της Μεσογείου αλλά και με τους όλους συναδέλφους πέρα τη Μεσογείου και γίνεται συνεργασία επιτακτικής βάσης. Έχουμε ποσότητα πληροφοριών. Ίσως μην το ξέρει και ο Σκάντη. Τεράστια ποιότητα των στοιχείων και η ποιότητα. Και η ποσότητα και η ποιότητα. Δεν χρησιμοποιούνται πάντα. Εκείνος που πρέπει να προτείνει κάτι και να συντάξει βιοοικονομικά μοντέλα και διαχειριστικά σχέδια δεν κάνει άλλο παρά να χρησιμοποιεί αυτή την κληρονομιά που είναι τεράστια. Τούτου λεχθέντος, όπως το είπα και στην παρέμβασή μου, σήμερα στη Μεσόγειο παράγονται οικονομικά μοντέλα μεγαλύτερης περιπλοκότητας εν συγκρίση με τη Βόρεια Θάλασσα όπου τα μοντέλα βασίζονται σε, σε αποθέματα ενός είδους. Στη Μεσόγειο βιοοικονομικά μοντέλα βασίζονται σε πολλαπλά είδη και είναι πολύ πιο περίπλοκα. Αυτό κατέστη δυνατόν χάρη στο γεγονός ότι υπάρχει επίπεδο πληροφοριών πολύ ψηλό. Πολλά, πολλές πληροφορίες. Πέραν αυτού, ο πρόσφατος κανονισμός για τη συλλογή στοιχείων του 2000 οδήγησε και σε άλλη πρόθεση για ανάπτυξη οικονομικών, επιστημονικών, κοινωνικών στοιχείων που πριν ήταν άγνωστα. Αυτό οδήγησε σε ωφέλη για τους εργαζομένους, αυτούς που απασχολούνται με την κατεργασία πιο σύγχρονου συστήματος ε, διαχείρισης της αλίας. Ευχαριστώ, κύριος Ντέιβις το ερώτημα, ευγνώμων είμαι τη πληροφορία. Το θέμα είναι τι γίνεται με τα αποθέματα. Ποια είναι η κατάσταση των αποθεμάτων, ήταν το ερώτημά μου, λέει ο κ. Ντέιβι. Δεν νομίζω ότι μου δόθηκε απάντηση σε αυτό. Αν είναι γνωστό, ένα από του τρει μπορεί να απαντήσει. Ο κ. Σπανιόλο. Ήδη απάντησα, νομίζω, εν μέρη. Υπάρχουν πολλαπλές ιδιαιτερότητες Στη Μεσόγειο δεν μπορούμε να κάνουμε stock assessment επί 150-200 ειδών. Τα βασικά είδη που είναι πάνω από το 60% των αποθεμάτων κανονικά κάνουν, είναι αντικείμενο stock assessment, αξιολόγηση. Θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη αξιολόγηση των, ε, των αξιολογήσεων που έκαναν οι αρμόδιοι φορεί Αποτίμηση. Ε. Για το θέμα αυτό, πάντα στην Επιτροπή για τη Μεσόγειο το συμπέρασμα το οποίο αντλείτο το για τα είδη μεγάλου βάθους υπάρχει υπεραλίευση. Τώρα η αλευτική προσπάθεια έχει μειωθεί πρόσφατα και θεωρητικά θα πρέπει να είχαν ε, μειωθεί οι αλλιεύσεις αυτών των ειδών. Αν είναι υπερβολική ή όχι η αλίευση ακόμα δεν μπορώ να το απαντήσω. Ίσως να υπάρχει πλήρης αλίευση ή υπεραλίευση. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ταχεία ανάκαμψη δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει τουλάχιστον πλήρης αλίευση αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν αλλάξει λοιπόν δραστικά τα πράγματα, αλλά περιμένω ανοιχτός, παραμένω ανοιχτός σε σχόλια και διορθώσεις από άλλους συναδέλφους. Ωραία. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Μπορούμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε και πάλι τους εισηγητές μας, τους ομιλητές μας σήμερα για τις πληροφορίες τους και δεν έχουμε κλείσει ακόμα. Τους αποχαιρετούμε. Μας μένει μονάχα ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη και οι συντονιστές έχουν ήδη κάνει έχει ήδη υπάρξει μια σύνοψη των ε, συμπερασμάτων των συντονιστών. Μπορούμε να την εγκρίνουμε αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Αυτά εργαστήκαμε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ όλους και τους διερμηνείς και τους βουλευτές οι οποίοι είναι παρόντες και λυπάμαι που δεν ήταν περισσότεροι. Και εδώ πρέπει να κάνουμε κάτι. Ευχαριστώ πολύ.